Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Ελέγχου Προϋπολογισμού και σας καλωσορίζω. Θα προχωρήσουμε κατευθείαν εις ε, την σημερινή ημερήσια διάταξη ε, εάν ε, το μικρόφωνο δεν δουλεύει, πέστε μου το, όχι δουλεύει. Λοιπόν, ε, Υπάρχουν ίσως επιθυμίες για αλλαγή της ημερησίας διατάξεως, όχι, οπότε ερχόμαστε στο πρώτο θέμα που είναι η έκθεση σχετικά με το ταξίδι στη Λιθουανία διότι εδώ επιληροφορηθήκαμε ε, για το υπόβαθρο της εκθέσεως Μαρινέσκου και για την ε, κατάργηση ε, και απενεργοποίηση του προηγουμένου πυρηνικού εργοστασίου Ιγναλίνα έχετε την έκθεση της αποστολής μπορέσαμε να διαπιστώσουμε επιτόπου ότι οι ε, διαμάχες οι οποίες ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αυτό δυστυχώς δεν έχουν ακόμη επιληθεί και ο στόχος της δικιάς μας εργασίας ήταν ε, βάσει της εκθέσεως του ελεγκτικού συνεδρίου να μπορέσουμε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Δηλαδή υπάρχει συμφέρον και των Λιθουανών πολιτών και δεν υπάρχει ε, σύγκρουση μεταξύ των Λιθουανών πολιτών και των υπολείπων πολιτών της Ευρώπης. Απλούστατα πρέπει να καταργηθεί και ε, να απενεργοποιηθεί σωστά αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο. Υπάρχει και η ε, έκτακτη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που λέει ότι ο φορολογούμενος ε, χρεώνεται 650.000 ευρώ αλλά η μέρα καθυστέρησες και ε, ο στόχος ο δικός μας ήταν να μπορέσουμε να υπάρξει μία οικονομική ε, πορεία των εργασιών αυτών και στο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπρεπε αυτό να τονιστεί. Αυτό είναι άλλωστε και ο στόχος του, της εκθέσεως αυτής. Ζητούμε από όλους τους συμμετέχοντες την ε, κυβέρνηση της Λιθουανίας και την εταιρεία Λιθουανία Power να ε, συμμετάσχουν και να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. Το δε μήνυμα ε, έφτασε σε εμένα σαν επικεφαλής της αντιπροσωπείας για να σας πω ότι από τη σκοπιά της κυβέρνησης της Λιθουανίας ε, οι αριθμοί που είχε υποβάλει η γραμματεία για την κατάρτιση της εκθέσεως δεν θεωρήθηκαν πλήρεις Είχαμε συλλέξει τα στοιχεία αυτά από επίσημες πηγές και ε, έχω ε, ασχοληθεί και με, ε, με το θέμα προσωπικά και είπα στην κυβέρνηση και στους ενδιαφερόμενους ότι κανείς δεν έχει συμφέρον να μην είναι σωστοί οι αριθμοί και θα πρέπει τα στοιχεία μας να προσαρμοστούν. Νομίζω όμως ότι ο υπεύθυνο για την ε, ε, κέντρωση των αριθμών αυτών δεν είναι η Επιτροπή μας αλλά αυτοί οι οποίοι συλλέγουν ε, τα στοιχεία και πρέπει να μας δίδουν τα σωστά στοιχεία εξού και πριν προχωρήσω στη συζήτηση θα ήθελα να δώσω τη την δυνατότητα στους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τοποθετηθούν και να μας πούν κατά πόσον οι αριθμοί οι οποίοι περιλαμβάνονται στην έκθεσή μας είναι σωστοί ή χρειάζεται ε, να ε, συμπληρωθούν και θέλω να καταλήξω με μία σαφή επισήμανση. Θέλουμε να στείλουμε μία ένδειξη ε, με τα ταξίδια των αντιπροσωπιών ότι τα προβλήματα θα λύνονται. Ε, δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να αποφασίσουμε σε ποιο συγκεκριμένο σημείο κάποιος έχει δίκιο ή αδικό. Αυτό γίνεται ε, στο Κοινοβούλιο μέσω του δημοσιονομικού ελέγχου και έτσι μπορούμε να πιέσουμε ε, την κυβέρνηση της Λιθουανίας να καταρτήσει ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει και τους συμμετέχοντες να μας ε, δώσουν σωστά αποτελέσματα διότι υπάρχουν και άλλα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λύθηκαν τέτοια προβλήματα γιατί όχι λοιπόν στη Λιθουανία προς κοινό συμφέρον. Πιστεύω ότι εδώ ψάχνουμε ε, ένα συμβιβασμό, μία λύση, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και αυτό θέλω να τονίσω και ε, να το περιλάβω και στα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τώρα τον ομόλογό μου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πει αν έχει κάτι επ' αυτού ε, και ενδεχομένως όποιος ε, παρέμβει μπορεί να μας πει εάν τα στοιχεία τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει ή η βάση των δεδομένων χρειάζεται να συμπληρωθεί και αν μπορείτε να σχολιάσετε την κατάσταση γενικότερα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρία σχόλια. Πρώτον, για τους αριθμούς που αναφέρονται εδώ για τα επενδυτικά προγράμματα. Σωστή είναι. Η άλλη δε αριθμή της έκθεσης από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω έχουν προκύψει από κάποια άλλη παρουσίαση. Είναι και αυτοί σωστοί αλλά δεν καλύπτουν τα πάντα. Διαβάζοντας την έκθεση δηλαδή μπορεί κανείς να μην έχει την πλήρη εντύπωση που θα έπρεπε να έχει. Παραδείγματος χάρη. Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα στήριξης της Κομισιόν προβλέπει και τη συντήρηση των πυρηνικών σταθμών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί έχει και κοινωνικές επιπτώσεις. Άλλο θέμα πληροφόρησης για την κοινή ή μεικτή επιτροπή που αναφέρεται με τη Λιθουανία. Αυτό είναι υποχρεωτικό από τη Συμφωνία Πλαίσιο. Δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, απλώς λειτουργεί μια κοινή διοικητική επιτροπή που συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο Δηλαδή συναντιόνται εκπρόσωποι της Λιθουανικής κυβέρνησης, της Κομισιόν της Τράπεζας και ορισμένοι άλλοι για να γίνεται κάθε φορά μια ανταλλαγή απόψεων για προβλήματα. Όσο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Β1, ο στόχος είναι όλα αυτά να συμπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015 ώστε να παροπληστεί ο πυρηνικός εκείνος σταθμός όσο δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Και λέει επίσης η έκθεση ότι η βασική συμφωνία θα μπορούσε να παγώσει ή να διακοπεί αν δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος μέχρι το τέλος Ιουλίου. Υπάρχει και ο δικός χάρτης προς τους δωρητές και την Κομισιόν για τις τεχνικές λύσεις που μπορεί να υπάρχουν και την επίτευξη συμφωνίας. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι όμως ότι ακόμα δεν έχουν γίνει τα βασικά και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση γιατί δεν έχουμε καμία ακόμη εγγύηση ότι ο δικός αυτός χάρτης πρόκειται πράγματι να οδηγήσει στην συμπλήρωση, την επίτευξη αυτού του προγράμματος μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε και τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής Ευχαριστώ. Ήμουν στη Λιθουανία και με ε, εξέπληξε και με ενόχλησε ε, και ε, δεν είναι δυνατόν να καίει κανείς τόσα πολλά χρήματα επί χρόνια. Και τώρα σταμάτησε το πρόγραμμα αυτό και ορισμένοι λέγουν δεν πειράζει για 30 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι πειράζει ε, ποιος ε, άρα ευθύνεται για αυτή την καθυστέρηση και τι θα γίνει με αυτή τη ζημία των 30 εκατομμυρίων ε, θα αποδοθούν στους φορολογούμενους και θα τους πούμε χάσατε λυπούμαστε ή θα αναλάβει κάποιος ευθύνες. Επίσης εντυπωσιάστηκα με την την ε, αντιμετώπιση των ανθρώπων. Δεν πρέπει να επιτρέπεται ε, ε, να δουλεύουν άνθρωποι με αυτές τις αντιλήψεις διότι νομίζω ότι οι νέες δημοσιονομικές συνθήκες συζητούνται στην Επιτροπή Ήτρε. Πόσο είναι βιώσιμο αυτό το οποίο συζητείτε, τι θα γίνει με το roadmap και τι θα γίνει αν δεν πετύχει πάλι. Δηλαδή, καταρχήν ποιος ευθύνεται ε, για την ε, καθυστέρηση και πώς θα κατανεμηθούν αυτά και πού θα αποδοθούν τα 30 εκατομμύρια, ε, τι θα γίνει και δεν χρειάζεται μία νέα οργανωτική δομή διότι πολλοί ε, συμμετέχοντες μας ε, είπαν ε, ότι μία ουδέτερη διατρησία θα ήταν η πιο ενδιαφέρουσα αλλά αυτά δεν θα θέλει, αυτή δεν θα θέλει να παρατείνει αυτή τη διαδικασία για να κερδίζει. Οπότε πώς θα αντεπεξέλθουμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση και μία παρατήρηση για τις τροπολογίες των δύο Λιθουανών ε, συναδέλφων καταρχήν όταν δεν ε, συμμετέχει κανείς ε, στην αποστολή δεν δικαιούται να κάνει παρατηρήσεις για την έκθεση της αποστολής. Δεύτερον αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα αλλά πρέπει μαζί με τους Λιθουανούς και όχι εναντίον τους να επιζητήσουμε μία λύση. Γι' αυτά είχα να πω σχετικά με το ταξίδι τις αντιπροσωπείες. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψή σας στη Λιθουανία. Σήμερα δεν ομιλώ ως εκπρόσωπος της χώρας αυτής, αλλά ως Ευρωβουλευτής που εκπροσωπεί το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, επειδή έχω ζήσει και εργαστεί στη Λιθουανία, έχω περισσότερες ίσως πληροφορίες από τις, για τις ισχύουσες διαδικασίες από άλλους. Σωστό είναι ότι η έκθεση αυτή δεν καλύπτει όλους τους αριθμούς και τις διαδικασίες διότι υπάρχει κάποια ασάφεια ως προς το ποιες διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται και ποιες όχι και αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Ο, λόγο, ο ρόλος της Μπέρτ καταρχήν είχε αποφασιστεί να παροπλιστεί εκείνος ο πυρηνικός σταθμός και να δοθούν ορισμένα χρήματα για αυτό το σκοπό στη Λιθουανία με τον όρο επειδή η Λιθουανία δεν είχε καμία τέτοια ανάλογη εμπειρία η χρηματική αυτή βοήθεια να χορηγηθεί μέσω της BERD και τώρα όλες οι πληρωμές από εκεί περνάνε. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν δικαιολογήθηκαν πλήρως με αποδείξεις και έγινε διαγωνισμός και η εταιρεία που κέρδισε το διαγωνισμό θα εφαρμόσει το πρόγραμμα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Λιθουανία ως χώρα μόνο την τεχνική επίβλεψη έχει αναλάβει ώστε να διασφαλίσει ότι η εταιρεία που κέρδισε το διαγωνισμό που ανέλαβε το πρόγραμμα δηλαδή θα εφαρμόσει όντως ό,τι προβλέπει το συμβόλαιο με βάση τις διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί από εκείνο. Αν λοιπόν το γενικό αυτό συμβόλαιο προβλέπει ορισμένες εγκαταστάσεις που θεωρούνται αμφίβολης ασφαλείας να παροπληστούν τότε πρέπει να πράξει ακριβώς αυτό ό,τι λέει το Συμβούλιο και αυτό να το επιτηρεί ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Υπάρχει μια υπηρεσία επιθεώρησης θεμάτων πυρηνικής ασφαλείας στη Λιθουανία και αυτή θα διασφαλίσει ότι όντως όλα γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια. Αυτό το λέω για να απαντήσω στο κατά πόσον υπάρχουν λόγοι σοβαρών και δικαιολογημένων αμφιβολιών. Εάν αποφασιστεί ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται αυτού του είδους τα containers ή οι εγκαταστάσεις αυτές είναι αμφιβόλου ασφαλείας θα, δεν θα χρησιμοποιηθούν. Ας μην επιστρέφουμε συνέχεια στις τεχνικές λεπτομέρειες. Πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα και για το μέλλον ποια ακριβώς είναι η ευθύνη του κάθε συμπαλόμενου μέρους και των αρμοδίων της Ένωσης. Συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε λοιπόν τίθεται το ερώτημα. Πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο γιατί κάθε φορά και σήμερα και ποιος θα είναι αύριο. Η ειδική πρόγραμμα είναι σωστό, αλλά η Λιθουανία δεν μπορεί να αποφασίσει από μόνη της ως χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αναζητήσουμε την τρίτη εναλλακτική συμβιβαστική λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι πρόσφατο, είναι πολλά χρόνια που τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Χωρίς να επανερχόμαστε συνεχώς στο παρελθόν γιατί αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος συνάδελφος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να προωθήσουμε ένα πρόγραμμα ε, και βρήκαμε ένα πολύ περίπλοκο πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί στην Λιθουανία και αυτή η περιπλοκή δεν προσφέρεται για να μας διευκολύνει ε, ούτε για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε ορισμένα θέματα ε, ούτε μεταξύ εθνικών αρχών αλλά ακόμη λιγότερο μεταξύ εθνικών αρχών, διεθνών αρχών, ε, Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας, ομολόγους και στις διαπραγματεύσεις και τα λοιπά να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό και θα έπρεπε να πούμε πολύ σαφώς ότι ε, εφόσον ε, ενδιαφερόμαστε πρέπει να πείσουμε και να πιέσουμε την κυβέρνηση της Λιθουανίας ότι αυτά που κάνει ε, θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και των πολιτών του και των γειτόνων του Βεβαίως ε, είναι πολύ άσχημη η διάθεση ε, των ε, ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό το εργοστάσιο. Είναι περήφανοι για αυτό, πιστεύουν ότι έχουν κάνει σωστή δουλειά και δεν ενθουσιάζονται όταν σκέφτονται ότι κάποιος έρχεται και τους λένε δεν μας αρέσει αυτό που κατασκευάσατε, κλείστε το. Εγώ έρχομαι από την περιοχή της Ρούρ, στη Γερμανία και έχουμε πουλήσει εργοστάσια στην Κίνα και ούτω καθεξής δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες αλλά ξέρω κοινωνιολογικά πόσο δυσάρεστη είναι η διαδικασία ε, της, ε, ε, του κλεισίματος ενός τέτοιου εργοστασίου. Πρέπει όμως να δώσουμε το μήνυμα ότι αυτό δεν έχει σχέση με μας και δεν πρέπει κανείς εδώ να παίρνει θέσεις υπέρ ή κατά απλούστατα πρέπει να, ε, να υπενθυμίσουμε τις υποχρεώσεις ε, τους στους ομολόγους μας διότι υπάρχουν Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και ε, ε, ε, φορολογούμενοι Ευρωπαίοι είναι και οι Λιθουανοί άρα να τους το επενθυμίσουμε με τον συνάδελφο Βέσλερ συμφωνώ ο συνάδελφος μάλλον με τη συνάδελφο Γκρέσλε συμφωνώ, ο κύριος Μπαλσίτης μας ε, ε, παρουσίασε την κάπως διαφορετική οπτική γωνία του και νομίζω ότι θα κινηθούμε ε, ειλικρινά και δίκαια αν ε, από τη μία πλευρά αντιμετωπίσουμε την Λιθουανική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας και τις επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά που πρέπει να αναλάβουν τις εργασίες της ε, ε, απενεργοποίησης του εργοστασίου και είπαμε ότι αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο πλευρών δεν μπορέσαμε να τη διατηρήσουμε διαπιστώσουμε κατά την αποστολή, δεν έχουμε τις γνώσεις, αλλά κάποιος πρέπει να προβεί σε αυτό το διαχωρισμό και να δρομολογήσει τη διαδικασία κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσει να αποδομηθεί ε, το εργοστάσιο και να υπάρχει δυνατότητα αυτό να υλοποιηθεί για να αποφύγουμε τις περαιτέρω καθυστερήσεις οι οποίες διαπιστώνονται. Μέσα στο πλαίσιο αυτό ίσως πρέπει να ενημερώσουμε τι έγινε με την αντιπροσωπεία και θα ήθελα τώρα η Επιτροπή ε, είτε εδώ προφορικά είτε γραπτά να μας πει τι έχει αμυφθεί από όταν ε, ε, πήγαμε στην Λιθουανία διότι ήρθε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στο Βίλνι για να προσπαθήσει να προωθήσει το θέμα. Ε, παρακολούθησα και στα μέσα ενημέρωσης στην συνέχεια την ε, κατάσταση αλλά καλό θα ήταν να έχουμε μία ενημέρωση είτε προφορική είτε γραπτή εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι καλό είναι να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα αλλά το, το, να μην έχουμε ένα μηχανισμό με τον οποίο θα υλοποιήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα σημαίνει ότι ε, ότι τα πράγματα δεν θα προχωρήσουν όπως τα έχουμε φανταστεί και προγραμματίσει. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέραν από αυτά τα οποία διαπιστώσαμε στην Λιθουανία για να εξασφαλίσει ότι προχωράει ο χάρτης πορείας και θα σεβαστώ αυτό ο το χάρτη πορείας εάν διαπιστώσω ότι υπάρχουν νέα μέσα ότι θα επιληθούν οι διαφορές διότι αν δεν υπάρχουν αυτά τα μέσα τότε δεν εξηγείται η αισιοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές και μπορείτε να τις απαντήσετε και στη συνέχεια μπορείτε να συμπληρώσετε με μία γραπτή δήλωση αν θέλετε. Ναι, φυσικά θα στείλουμε γραπτή, θα υποβάλουμε γραπτή απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα αν το δέχεστε, αν δεν έχετε αντίρρηση. Το θέμα είναι, μπορείτε σήμερα να απαντήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα ερωτήματα. Ένα σύντομο σχόλιο μπορώ να κάνω και μετά θα τα αναφέρουν οι γραπτές απαντήσεις λεπτομερέστερα. Λοιπόν, για το ποιος είναι υπεύθυνο. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Έχουμε ακόμη δυσκολίες και αυτό οφείλεται στο ότι δεν είναι άσπρο μαύρο. Υπάρχουν ευθύνες και από τις δύο πλευρές και πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν προσπάθειες να βρεθεί μια λύση. Και όταν λέω οι δύο πλευρές εννοώ τον εργολάβο και τον εργοδότη Πρέπει το συμβόλαιο να εφαρμοστεί ακριβώς όπως αναφέρεται και πρέπει το IPP να φροντίσει για την εφαρμογή. Και στη συνέχεια πρέπει να δοθεί και η άδεια. Τώρα για τα 30 εκατομμύρια δεν μπορώ να σχολιάσω, δεν γνώριζα αυτόν τον αριθμό. Uh, Για το άλλο θέμα, εντάξει, το ξέραμε. Αλλά επίσης ξέραμε ότι χρειάστηκε να αλλάξει η εργοληπτική εταιρεία της κατασκευής εκεί και γι' αυτό καθυστέρησε χρονικά. Τώρα, τι έκανε η Κομισιόν από τον Ιούλιο εφάρμοσε την απόφαση της διάσκεψης των δωρητών του Ιουνίου. Δηλαδή μαζί με την Baird που θα έκανε την, ε, θα χορηγούσε τις πληρωμές στείλαμε μία επιστολή στο INPP όπου ζητούσαμε περαιτέρω πληροφορίες για τη συνέχεια και ο διευθυντής Πίτερ Φάρος είχε πάει στη Λιθουανία λίγες μέρες μετά τη δική σας συνεδρία και θα ξαναπάει την επόμενη εβδομάδα στην τράπεζα για να συζητήσει με όλους τους υπεύθυνους και αρμόδιους. Και το INPP θα απαντήσει στους δωρητές και στην Κομισιόν και τότε θα έχουμε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία μπροστά μας για να δούμε αν πρέπει να διακοπεί ή όχι η χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο και μετά πρέπει να μιλήσουμε για τη συνέχεια της διαδικασίας γιατί εδώ βιαζόμαστε. Ευχαριστώ. Έχω δύο επιπρόσθετες ερωτήσεις για γραπτή απάντηση. Ε, όταν λέτε ότι δεν γνωρίζετε τα 30 εκατομμύρια αυτά, ε, είναι από τους αριθμούς που μας δόθησαν 1000 ευρώ το μήνα και σε τέσσερα χρόνια είναι ακόμη περισσότερα. Και αν εσείς δεν γνωρίζετε το ποσό των 30 εκατομμυρίων, ότι είναι οι αριθμοί με ε, τους οποίους έχετε για το κόστος των ε, καθυστερήσεων και ποιος είναι ο authorizing officer για αυτά τα θέματα, ο κύριος Μπαλτσίτης. Όπως είπε και η συνάδελφος Ινκεμπουργκ Γκλέσλερ, δεν έχω, δεν μπορεί κανείς να προσθέσει πολλά το κυριότερο θέμα είναι ποιος είναι ο υπεύθυνο αυτού του τεραστίου προγράμματος που δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Να ζητήσω κάτι. Η Κομισιόν θα ήθελα να μας υποβάλει ένα έγγραφο που να αναφέρει τις ευθύνες, τις συγκεκριμένες ευθύνες της Μπέρντ της Νιούκομ γιατί υπάρχουν όροι που προβλέπονται στο συμβόλο που δεν είναι τίποτα μυστικό και θα ήθελα να μας τα πει. Ο εκπρόσωπος μάλιστα της Κομισιόν μπορεί να μας πει αν έχουν δίκιο οι εκπρόσωποι της Λιθουανίας που ζητούν πρόσθετα έγγραφα εάν ο εργολάβος δεν έχει εφαρμόσει το συμβόλαιο που Ωραία. Αυτά είναι πρόσθετα ερωτήματα. Θέλετε να σας τα πει τώρα η Κομισιόν. Σύντομα ή τώρα και πιο λεπτομερώς γραπτά. Ναι, ένα σχόλιο για την πρόσθετη τεκμηρίωση. Εδώ προβλέπονται όλα αυτά. Η τεκμηρίωση προβλέπεται ώστε μετά την κατασκευή να δοθεί η άδεια λειτουργίας και δεν είναι τίποτα καινούριο, όλα αυτά τα λέει το συμβόλαιο. Και ο Λιθουανός ρυθμιστής τα ξέρει. Τα υπόλοιπα γραπτός. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τελειώνει αυτή η συζήτηση εδώ με την πρόταση η σύσταση του συναδέλφου Μπαλτσίτης που ήταν μέλος και της αντιπροσωπείας που πήγε εκεί να συμπεριληφθεί και να συζητηθεί μεταξύ ομάδων για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε καμία συνένεση ή συμβιβασμό και να λήξει τελικά η συζήτηση μετά την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 να αναφέρω ότι πρόκειται για μια περίπτωση, θα έλεγα, θεσμικής ανοριμότητας που ξεπερνάει το Κοινοβούλιο σε άλλες ε, καταστάσεις, σε άλλες συγκυρίες μέσα από την ε, Συμβουλευτική Επιτροπή. Σήμερα με την απαλλαγή του προϋπολογισμού αυτή η συμφωνία κυρίων του 70 είναι ξεπερασμένη και αυτό φάνηκε. Δεν θα έπρεπε να δεχτούμε λοιπόν να επανέλθουμε σε αυτήν τη συμφωνία κυρίων. Γιατί το 2000 ε, και υπό η Ισπανική Προεδρία με σοσιαλιστική κυβέρνηση το Συμβούλιο είχε δεχτεί αυτή η περίφημη, ότι αυτή η περίφημη συμφωνία κυρίων έπρεπε να ξεχαστεί ότι ήταν ένα μέσο που δεν είναι καθόλου επίκαιρο και συμβατώ με την ε, θεσμική οριμότητα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι να προχωρήσουμε. Εμείς έχουμε μπροστά μας ένα θέμα καθαρά θεσμικό. Πρόκειται για μία μάχη πολιτικοθεσμική, περισσότερο από ότι μία μάχη ελέγχου προϋπολογισμού, διότι ο διοικητικός ε, προϋπολογισμός του Συμβουλίου είναι αμεληταίος ε, αν τον συγκρίνουμε με τον ε, γενικό προϋπολογισμό. Και για την Επιτροπή μας επίσης, αλλά είναι όμως πολύ σημαντικό από θεσμικής πλευράς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εγώ ως εισηγήτρια θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το παραγωνίσουμε σε μία μόνιμη άρνηση και αποσιώπηση για λόγους ευκολίας. Εγώ θεωρώ και χαιρετίζω ότι αυτό, αυτό το σεμινάριο που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να πείσουμε και το άλλο θεσμικό όργανο που παραμένει αμετάκλητο σε αυτήν την ανοριμότητα και στην απόρριψη. Όλος ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να είναι ελεγμένος και να είναι υπόλογος έναντι στο κοινοβούλιο. Και δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πλάγιες εξόδους και παραθυράκια. Εμείς από το 2000 και μετά έχουμε μια κατάσταση ιδιαίτερα πολύπλοκη. Η Επιτροπή μας προσπάθησε να εργαστεί για να δει πώς θα μπορούσε να μετακινήσει την ε, βούληση, να αλλάξει τη βούληση του Συμβουλίου. Στο παρελθόν δεν είχαν έτσι τα πράγματα. Αυτή η θεσμική συμφωνία θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα θεσμικά όργανα και θα πρέπει να προετοιμαστεί από την Κοκομπού και το Κοινοβούλιο παρά τις ορισμένες επιφυλάξεις αποφάσισε η Επιτροπή αυτή πέρα από την ετήσια απαλλαγή να βρει μία, έναν τρόπο προσέγγισης του, του Συμβουλίου. Αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας στο τραπέζι και είναι το ρίσκο είναι να υπάρξει πάλι άρνηση του Συμβουλίου και αυτό χωρίς επιπτώσεις. Εκτός αν καταφέρουμε να βρούμε κάτι το εφάνταστο και καινοτόμο και κινηθούμε πολιτικά. Στην πολιτική μάχη που πρέπει να δώσουμε. Εκείνο το οποίο πρέπει να αποφύγουμε είναι να προσφύγει στο δικαστήριο το Συμβούλιο, πράγμα που δεν έκανε μέχρι τώρα γιατί δεν το ενδιέφερε. Η άλλη περίπτωση είναι να, να, πάμε κι εμείς να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Αυτό όμως θα οδηγούσε σε μία παράλυση στην όλη διαδικασία της απαλλαγής. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι κίνδυνοι. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να μας το ξεκαθαρίσει αυτό. Μια άλλη διέξοδος θα ήταν να δεχθούμε την πρόταση του Συμβουλίου. Δηλαδή, δεδομένου ότι η συνθήκη προβλέπει απαλλαγή προς την Κομισιόν, εφόσον δίνουμε απαλλαγή στην Κομισιόν, καλύπτουμε έτσι και την απαλλαγή στις διοικητικές δαπάνες του Συμβουλίου. Υπάρχουν συνάδελφοι που σκέφτηκαν και αυτή τη λύση. Εγώ πιστεύω όμως ότι σε αυτό το σεμινάριο θα έπρεπε να συζητήσουμε και αυτή την πιθανότητα και τους κινδύνους που ενηχεύει. οι συνάδελφοι πρότειναν ε, μια μαξιμαλιστική θέση, δηλαδή αφού το Συμβούλιο δεν δέχεται την απαλλαγή, τότε θα απαλλάξουμε την Κομισιόν. Όμως, όταν αναφέραμε εμείς πολλές φορές τον Επίτροπο Σεμέτα τον κίνδυνο της έλλειψης συνεργασίας, Μα είπε ότι αν δεχόμασταν την πρόταση του Συμβουλίου τότε θα ήταν η Κομισιόν που θα το αναλάμπανε το θέμα. Υπάρχουν όμω και άλλε λύσεις. Η περίφημη εθνική δήλωση για τις δαπάνες των κρατών μελών. Δεν ξέρω στο Συμβούλιο τι άλλη φόρμουλα μπορούμε να βρούμε. Επίσης υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα ένα μνημόνιο που θα, είναι βάση μιας, θα αποτελέσει βάση μιας θεσμικής συμφωνίας και όπου θα διαπιστώσουμε εμείς ποιοι είναι οι διαφορετικοί ρόλοι και σε τι υφίστανται αυτοί οι ρόλοι. Διότι σε περίπτωση απαλλαγής η συνθήκη προβλέπει διαφορετικούς ρόλους. Η Κομισιόν προτείνει, το Κοινοβούλιο αποφασίζει και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και τον κορμό μιας μελλοντικής συμφωνίας. Και σε αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει το σημερινό σεμινάριο. Εγώ σήμερα ε, το πρωί που πήρα τα έγγραφα δεν διαπίστωσα καμία αναφορά των εμπειρογνωμόνων για αυτό το βασικό μνημόνιο για να μπορέσουμε να έχουμε μία συμφωνία. όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η μάχη, κοινοβούλιο, συμβούλιο, έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο, ένα άλλο πεδίο μάχης, που είναι η μάχη των ε, ε, δημοσιονομικών προπτικών 2014-2020. Η δικιά μας η μάχη είναι ε, πλευρική μάχη. Αλλά επειδή εγώ είμαι σκληροκέφαλη, γιατί είμαι από την Αραγωνία και από σκληροκεφαλιά στην Αραγωνία δεν χάνουμε ποτέ μάχες, θα επιμείνω. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο χρειάζεται να υπάρχει και η υπεποίθηση σε αυτήν την Επιτροπή ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε αυτή τη θεσμική σχέση στο πλαίσιο της απαλλαγής, πρέπει να αναγνωρίσουμε τον καθοριστικό ρόλο του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο πρέπει να έρθει να συζητήσει, να συνδιαλλαγεί και να σταματήσει αυτή η φόρμουλα έστειλα μια, ένα γράμμα και άντε να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να έρθουν εδώ και να, να εργαστούμε σοβαρά και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα θεσμικής ανοριμότητας. Εγώ δεν είμαι ούτε αθώα ούτε αφελής, ξέρω ότι υπάρχει πολιτική δυσπιστία μεταξύ των δύο οργάνων, αυτό αποτελεί τμήμα της πολιτικής ανοριμότητας και αντί εμείς να χασκογελάμε κάθε φορά που απουσιάζει το Συμβούλιο όταν το προσκαλούμε, θα έλεγα ότι πρέπει να το πάρουμε πολύ πιο στα σοβαρά διότι οι κοινωνίες σε μια περίοδο κρίσης και δυσπιστίας έναντι των πολιτικών αρχών τέτοιου είδους συζητήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή αυτής της τάσης της δυσπιστίας δηλαδή. Δυσπιστεί το Συμβούλιο έναντι του Κοινοβουλίου γιατί, τι θεωρεί ότι και το κοινοβούλιο παίζει ρόλο σε αυτήν την δημιουργία δυσπιστίας και μια αυτοκριτική κακό δεν κάνει. Πρέπει να κοιτάξουμε να ξεπεράσουμε αυτήν τη θεσμική ανοριμότητα χωρίς βέβαια να γνωρούμε ότι υπάρχει αυτή η ευρύτερη μάχη που δίνεται για τις δημοσιονομικές προπτικές 14-20. Ε, εγώ είμαι αισιόδοξη, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ και εκφράζω την ικανοποίησή μου για αυτό το σεμινάριο και ελπίζω κύριε Πρόεδρε ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να δούμε τι λύσεις θα μπορούσαμε να προωθήσουμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι ανάξιο των πολιτών μας. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ για αυτή την πολύ ενθουσιώδη παρουσίαση. Βλέπετε ότι συζητήσαμε επανειλημμένων, συζητήσατε επανειλημμένως για ένα πεδίο μάχης. Ε, ελπίζω ότι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πεδία μάχης του παρελθόντος έχουν αντικατασταθεί ε, ένα έχουν αντικατασταθεί από ένα πεδίο όπου απλώς ξυφομαχούμε και τώρα δίνω το λόγο για την πρώτη παρουσίαση στον κύριο Ρώση και τον παρακαλώ να παρουσιάσει το θέμα του. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δώσατε να μπορέσω να μιλήσω εδώ, όχι μόνο ε, από πλευράς ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά διότι είμαι ειδικό στα θέματα του δημοσιονομικού ελέγχου και γι' αυτό αισθάνομαι ότι συμμετέχω. Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θα χαρίσω που θα μιλήσω εδώ, γιατί όποιος έχει διαβάσει το κείμενό μου θα γνωρίζει ήδη ότι δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου από, την, ε, από το πρωτογενές δίκαιο μία βάση ε, για την εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Βεβαίως ο συνάδελφός μου παρουσιάζει την αντίθετη θέση, αλλά εγώ ε, νομίζω ότι τα σχόλιά μου θα ενισχύσουν τη θέση του Συμβουλίου. Μιλώ εδώ σήμερα σαν ε, ε, νομικός βάσει του ισχύοντος δικαίου. Δηλαδή θα μιλήσω για το εάν υπάρχει αρμοδιότης απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι αν υπάρχει ανάγκη απαλλαγής πράγμα το οποίο μέσω του τροποποιημένου δικαίου του Λέγκα Φερέντα μπορεί ίσως να στηριχτεί ε, και ε, ε, δεν ξέρω ποια θα είναι η μελλοντική δομή της Ευρώπης το σημείο κινήσεως όπως είπε και η συγγήτρια αυτών των νομικών θεμάτων είναι το άρθρο 319 το, της συνθήκης όπου λέγεται ότι ε, το ε, ε, ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να απαλλάξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αυτό το κείμενο είναι τόσο σαφές που εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Άρα δεν βλέπω γιατί κανείς γιατί κανείς θεωρεί ότι το κοινοβούλιο πρέπει να απαλλάξει και το συμβούλιο. Ο μόνος ο οποίος είναι αποδέκτης της απαλλαγής είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό εξηγείται και ε, λειτουργικά διότι βλέπετε ότι στο παρελθόν μέχρι το 1970 ήταν ο οργανισμός ο οποίος απείλασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το 1977 ισχύει ο κανόνας που ισχύει ακόμη ότι το Κοινοβούλιο προβαίνει σε μία, ε, η Επιτροπή προβαίνει σε μία σύσταση και αποφασίζει τελικά το Συμβούλιο προβλέπει, προβαίνει σε μία σύσταση και το Κοινοβούλιο απαλλάσσει. Αλλά στον πυρήνα της απαλλαγής βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι αυτό έχει σχέση με το άρθρο 317 της συνθήκης και σύμφωνα με τη διάταξη αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προπονομισμού άρα πρέπει να απαλλάξω τον υπεύθυνο σύμφωνα με την βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις ε, οπωσδήποτε τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απαλλάσσεται και δεν βλέπουμε αν πρέπει να απαλλαγούν και άλλοι. Εγώ δεν ε, ακολουθώ αυτό το σκεπτικό διότι τότε θα μπορούμε να ρωτήσουμε μήπως θα έπρεπε να απαλλαχούν και τα κράτη-μέλη ή ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία απαλλάσσει άλλα θεσμικά όργανα ή άλλα άτομα δηλαδή αν θα υπάρχουν και άλλοι αποδέκτες της απαλλαγής αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά παρακάμπτουν ιστορικά το το θέμα και δεν ε, έχουν νομική βάση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποτελούν από κοινού την νομοθετική αρχή και πρέπει ε, να να λυθεί το θέμα διότι ε, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες το 2014 αναγνωρίζονται και επισήμως νομικά ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σαν ε, αρχές νομοθετικές αλλά το να θεωρηθεί ότι ε, άλλαξε θέση το κοινοβούλιο και από ε, υπεύθυνο να απαλλάξει ε, πρέπει να γίνει υπεύθυνο να απαλλαγεί δεν με βρίσκει σύμφωνο διότι τότε δεν υπάρχουν πλέον ευθύνες και αυτό το λέω με κάθε σεβασμό προς τις αντίθετες απόψεις διότι είναι σαν να ζητάτε να ζητά το κοινοβούλιο να απαλλαχθεί μόνο του πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην δώσει απαλλαγή στον εαυτό του διότι ορισμένοι ευρωβουλευτές διαφωνούν ε, δηλαδή όλες οι άλλες αποφάσεις απαλλαγής θα ήταν ε, παρακινδυνευμένες και έχουν μόνο τον χαρακτήρα χαρακτήρα κάποιας διακήρυξης απόψεων. Ε, νομικά λοιπόν και όχι πολιτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται ε, σύμφωνα με ε, το νόμο το, οι συνθήκες είναι το σύνταγμα οπότε δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει από αυτά διότι ε, δεν μπορούμε να την ε, λύσουμε διότι ε, το 2007, 9, 12 μπορείτε να έχετε αντίθετες απόψεις αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε το ισχύον δίκαιο. Θα μπορούσε να υπάρξει μια αλλαγή των συνθήκων αλλά είναι μια μακριά διαδικασία. Εδώ λοιπόν αυτό που πρέπει να κοιτάξω είναι ε, τι είναι συμπεφωνημένο ε, και από αυτό δεν μπορώ να αποκλείσω. Δεν ξέρω πώς ε, θα αντιμετωπίζει το θέμα ε, η νέα ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός ε, και εις βάρος της ε, διαφάνειας δεν μπόρεσα να βρω εις τον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή στο διαδίκτυο τον νέο προϋπολογισμό δηλαδή δεν έχω μπορέσει να βρω το σχέδιο του επομένου προϋπολογισμού και δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζω αντιμετωπίζετε το όλο θέμα από αυτή την οπτική γωνία. Ένα άλλο θέμα και εδώ δεν θα σας ευχαριστήσω είναι ότι κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως φέρει όλη την ευθύνη για την εκτέλεση ε, του, του προϋπολογισμού και αυτό λέγεται στο άρθρο 317 και ε, επίσης ε, δεν θα σκεφτείτε παραδείγματος χάρη για τη Λιθουανία ή για τη Γερμανία να αρνηθείτε απαλλαγή γιατί στις χώρες αυτές δεν έχει εκτελιστεί σωστά ο προπολογισμό. Ο αποδέκτης απαλλαγής είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το ίδιο συμβαίνει και με την κυβέρνηση σε ένα ε, κράτος μέλος και το ίδιο ισχύει και για, τους, τα άλλα θεσμικά όργανα. Εάν κάποιο θεσμικό όργανο δεν εκτελέσει σωστά τον προϋπολογισμό, ο υπεύθυνο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι το, η οργάνωση μέλος που εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, εάν λοιπόν θέλετε ε, να αρνηθείτε την απαλλαγή του προπολογισμού πρέπει να στρέφεστε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι στο Συμβούλιο και αυτό είναι λογικό μπορεί βέβαια να σας τρομάζει αλλά τώρα εδώ εμπλέκεται και η γερμανική μου υπηκότητα ε, που κατανοεί το ομοσπονδιακό κράτος Λοιπόν, σκεφτείτε, εάν αρνηθεί μπορεί το ε, Bundestag, το Ομοσπονδιακό, η Ομοσπονδιακή Βουλή να αρνηθεί ε, στην Ομοσπονδιακή Γερουσία την απαλλαγή, όχι βέβαια διότι το θέμα δεν είναι αν τα λάθη έχουν διαπραχθεί ή στον τομέα των δικών της δραστηριοτήτων ή των ε, διαφόρων υποδεστέρων οργανώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα κράτη-μέλη, διότι βεβαίως το ομοσπονδιακό ο ε, η Ομοσπονδιακή Βουλή μπορεί να αρνηθεί να απαλλάξει ε, το... τη Βουλή ενός κρατηδίου εάν δεν εκτελεστεί στο κρατήδιο αυτό σωστά ο ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Υπάρχει δηλαδή μία διαφορά και δεν μπορώ να αντιληφθώ τη θέση σας ε, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του εσωτερικού τομέα στον οποίο εκτελείται ο προϋπολογισμός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία είναι υπεύθυνη απέναντί σας και ε, η οποία ε, πρέπει να, ε, να προβληματιστεί για κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και στο άρθρο 319 έχουμε και ένα μέσων ε, για να το πράξουμε. Ε, φαντάζομαι ότι άλλοι έχουν διαφορετικές απόψεις αλλά εγώ νομίζω ότι βλέπουμε ε, ότι υπάρχει στην παράγραφο 1 η απόφαση απαλλαγής και μετά υπάρχουν οι παρατηρήσεις και τα μέσα με τα οποία μπορούν να υποβληθούν οι παρατηρήσεις και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τα παραλαμβάνει αυτές τις παρατηρήσεις πρέπει να προβεί στις διευκρινήσεις εάν υπάρχουν λάθη δομικά ή εάν υπάρχουν μεμονωμένα προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι μια επαρκής δρομή για να μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις διαφορές. Πρέπει να σας πω ότι ε, δεν ισχύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο, μόνο του φέρει την ευθύνη της ευρωπαϊκής νομιμοποίησης ε, και υπάρχουν ε, δύο πυλώνες. Ως εκ τούτου δεν θεωρείται το Συμβούλιο ενδεχομένως ε, σαν ε, δημοκρατικό όργανο και δεν μπορείτε να το προσβάλλετε διότι θα προσβάλλατε όλη την αρχιτεκτονική του οικοδομήματος της Ευρώπης αλλά θα πρέπει να παραμείνει η του υπολογισμού στην την ευθύνη του θεσμικού οργάνου που τον ε, εκτελεί. Ε, με ρώτησαν ε, τι έγινε το 1970, την πρώτη φορά δηλαδή που ένεπλακει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην απαλλαγή του προϋπολογισμού, οι οποίοι είπαν ότι δεν μπορεί να απαλλάξει το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ούτε τον εαυτό του και ε, τουλάχιστον ε, εάν χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της χώρας μου της Γερμανίας αλλά και της Αυστρίας ή και ε, των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός της Ευρώπης μπορούμε να δούμε ότι δεν μπορεί ένα κοινοβούλιο να απαλλάξει τον εαυτό του από την εκτέλεση του προπολογισμού του. Τώρα όμως ερχόμαστε σε ένα βασικό θέμα, σε μία διαφορά. Δηλαδή ε, το θέμα του τι, ποιον μπορείτε να απαλλάξετε αλλά και το θέμα το τι πληροφορίες χρειάζεστε και προφανώς ε, θα πρέπει η απόφασή σας να λαμβάνετε βάση πληροφοριών σωστών και γι' αυτό πρέπει να έχετε τις πληροφορίες και έτσι ερμηνεύω το άρθρο 319 το οποίο σας ε, δίνει δίνει τη δυνατότητα να ε, έχετε πληροφορίες και εξ και τις πληροφορίες αυτές θα τις ζητήσετε ε, από, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είτε παρακάμπτεται το δίκαιο είτε όχι ουσιαστικά οι πληροφορίες πρέπει να σας δίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι ε, διευκρινίζεται το οικοδόμημα μεταξύ των εσωτερικών δομών και εξωτερικών δομών όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που πρέπει να βρει, να συλλέξει και να σας μεταδώσει τις πληροφορίες. Τώρα, ε, όσον αφορά την σύσταση της ε, απαλλαγής, εάν πρέπει να βασιστείτε στις υπάρχουσες πληροφορίες, ε, αυτό θα το, θα το αρνηθώ, διότι εάν το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο πει δεν χρειάζομαι όλες αυτές τις πληροφορίες τότε δεν δεσμεύεστε και νομίζω ότι μπορώ εδώ να προσθέσω ότι στην ισχύουσα δομή ε, των θεσμικών οργάνων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο μόνος αποδέκτης ε, αιτήσεων για πληροφορίες. Δεν ήξερα ότι θα μιλούσαμε σήμερα και για το ε, ατομικό εργοστάσιο της Λιθουανίας αλλά εσείς μιλάτε για κρίση πράγμα το οποίο ίσως δεν αντιλαμβάνεται η ομίγυρης εκτός ε, κοινοβουλίου διότι ε, ο προϋπολογισμός διαχείρισης του Συμβουλίου δεν είναι τόσο εκτενής διότι ε, εκτός από δύο-τρεις εξαιρέσεις οι εργασίες δεν εκτελούνται από το Συμβούλιο άρα δεν βλέπω ποια είναι η αξία της απαλλαγής του. Ε, δεν, ε, δεν ερμηνεύω την πολιτική σκοπιά, σκοπιμότητα αλλά ε, εφόσον θέλει κανείς να ανταποκριθεί στην κρίση δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει και Τέλος, κυρία Σέντερ, το υπόμνημά σας ε, το έχω δώσει για μετάφραση και έτσι δεν το γνωρίζω ακόμη πλήρως. Με ενδιαφέρει όμως, θα προσπαθήσω στη συνέχεια να το εξετάσω. Νομίζω ότι οι προτάσεις σας είναι επικοδομητικές και τώρα ολοκληρώνω Νομίζω ότι είτε πρόκειται ε, για υπόμνημα είτε για διαθεσμική συμφωνία ε, δεν θα μπορέσουμε να παρακάμψουμε την ε, απαλλαγή οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να σεβαστούν τη διαδικασία αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορείτε να αρνηθείτε την απαλλαγή του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρώση. Όντως υπάρχουν πολλά ερωτήματα αλλά συμφωνήσαμε ότι καταρχήν θα ακούσουμε τις διάφορες απόψεις και θα δώσω τώρα το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια την κυρία Φλωρόν Σαλχέλ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και για μένα είναι τιμή να σας αναφέρω εδώ ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί είναι ουσιώδες για όλες μας τις κοινωνίες και την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, δηλαδή το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου, της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Έχω μια παρουσίαση PowerPoint Τέλος πάντων και χωρίς αυτό γίνεται. Άκουσα να γίνεται λόγος για τον Ευρωπαϊκό Λαό και για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον εκπροσωπεί. Αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα γιατί μίλησε ο προηγούμενος για τη γερμανική πραγματικότητα αλλά για τη γαλλική για την οποία θα ήθελα να αναφερθώ είναι ιδιαίτερα άγνωστο στοιχείο η δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη ενώ είναι η κεντρική ιδέα στην οποία θέλω εγώ να στηριχτώ εδώ. Πρέπει να δίνεται λόγος βέβαια για τη χρήση του προϋπολογισμού ακόμη και αν οι πολίτες άμεσα <clears throat> δεν έχουν στοιχεία για την χρήση αυτή. Ποια είναι η γενικότερη φιλοσοφία λοιπόν που θέλω να αναφέρω. Τα πράγματα είναι για μένα σαφή όπως θα έλεγε και ο προηγούμενος ομιλητής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η μοναδική αρχή δημοκρατικού ελέγχου στην Ένωση. Το Συμβούλιο δεν χαρακτηρίζεται με ένα από έλλειψη δημοκρατίας, αλλά δεν ασκεί αυτό τον δημοκρατικό έλεγχο. Έχει δικό του τρόπο λειτουργίας μέσω των κρατών μελών και των κυβερνήσεων του επόμενου γίνεται και εκεί ένας έμεσος δημοκρατικός έλεγχος. Λοιπόν, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται, το ξέρετε πολύ καλά, από τις εθνικές εισφορές και επομένως από τι αποτελείται από τους φόρους μας των πολιτών που βέβαια πληρώνονται εθνικά αλλά ισχύει ότι κάθε ευρώ που δαπανάται από, από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό όργανο πρέπει να μπορεί να δικαιολογείται και να ελέγχεται από την αρχή δημοκρατικού ελέγχου, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει όμως εδώ και χρόνια ένα πρόβλημα και είναι το θέμα μας σήμερα. Το Συμβούλιο δεν θέλει, δεν επιθυμεί να υποβάλει τα έγγραφα που συζητάει, ούτε απαντάει σε ερωτήσεις. Το Κοινοβούλιο πάντα ζητούσε μεγαλύτερη συνεργασία με το Συμβούλιο για να μπορέσει έτσι να ασκήσει πιο αποτελεσματικά και πιο διαφανώς τον έλεγχο της χρήσης του προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο αρνείται να κάνει πλήρως αυτή τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο εν ώψη και της απαλλαγής που πρέπει να χορηγεί το Κοινοβούλιο για το Συμβούλιο και τη Επιτροπή. Υπάρχουν λοιπόν εδώ διαφορετικές αναγνώσεις και ερμηνείες της συνθήκης. Θα καταλάβατε ήδη που θέλω να καταλήξω. Διαφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής ο κύριος Ρώση, ιδιαίτερα όμως από, με το ότι είναι όλα απριόρι καθαρά και εξάστερα. Και εγώ νομικός είμαι και ξέρω ότι υπάρχει η νομολογία του δικαστηρίου που δείχνει ότι δεν είναι όλα καθαρά και εξάστερα και διαφανή. Το 319 το ερμηνεύουν διαφορετικά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ενώ είναι ρητό. Για το Συμβούλιο η Κομισιόν είναι η αρχή θεματοφύλακας των συνθήκων, εκείνη ε, ασκεί τον προϋπολογισμό και όταν δίνεται απαλλαγή προς την Κομισιόν αυτό σημαίνει για το Συμβούλιο ότι δίνεται απαλλαγή προς όλα τα όργανα. Ενώ αντίθετα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι δεν μπορεί να ασκήσει πλήρως το καθήκον του δημοκρατικού ελέγχου παρά μόνο αν έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που του χρειάζονται. Και άρα τα έγγραφα του Συμβουλίου προς το οποίο συχνά ζητάει τεκμηρίωση και το οποίο του την αρνείται. Υπάρχουν λοιπόν δύο διαφορετικές ερμηνείες της συνθήκης εδώ. Το θέμα λοιπόν που θέτω είναι πώς μπορούμε να λύσουμε τη διαμάχη αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς του Συμβουλίου και στα έγγραφα που θα του ζητήσει και πρέπει την απαλλαγή που δίνει προς το Συμβούλιο να τη δίνει ειδικά γι' αυτό μεμονωμένα και θα σας το εξηγήσω. Να δούμε ποιο είναι το ίσχυον δίκαιο, είναι, ποια είναι τα καθήκοντα που επιβάλλει αλλά και ποιες ασάφειες μπορεί να υπάρχουν. Στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι η πρακτική, πώς ασκείται αυτό το δίκαιο και τέλος θα σας προτείνω και μερικές πιθανές λύσεις που σίγουρα δεν θα ικανοποιήσουν τους πάντες με την ανάλογη νομική επιχειρηματολογία. Λοιπόν, πρώτο, το 319 της συνθήκης, το άρθρο 319. Η διαφορετική του ερμηνεία δείχνει ότι περιέχει κάποια ασάφεια μας λένε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλάσσει την Επιτροπή την προτάση του Συμβουλίου και με την υποστήριξη του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτό δεν είναι καθαρό και εξάστερο για να επαναλάβω αυτά που είπατε εσείς προηγούμενοι ομιλητά. Τι θα πει η προτάση του Συμβουλίου. Αυτή η έκφραση υπονοεί ότι το Συμβούλιο είναι και αυτό αρχή ελέγχου του προϋπολογισμού. Αυτό δεν ισχύει. Δεύτερη ασάφεια. Το κείμενο βασίζεται στο ότι όπως λέει το Συμβούλιο η Κομισιόν είναι η μόνη αρχή χρήσης του προϋπολογισμού. Αλλά δεν ισχύει ούτε αυτό. Διότι τα πράγματα δείχνουν ότι η Κομισιόν πόρο απέχει από το να είναι η μόνη αρχή χρήσης του προϋπολογισμού αν θέλουμε να γίνει ένας πραγματικός έλεγχος και διαπιστώνουμε ότι δεν είναι η μόνη τέτοια αρμόδια αρχή Κομισιόν τα πράγματα είναι σαφή. Δηλαδή, κάθε όργανο που ασκεί που, τον προϋπολογισμό πρέπει να γίνεται αντικείμενο δημοκρατικού ελέγχου. Ο δημοσιονομικός κανονισμός, το άρθρο 50, λέει όντως ότι η Κομισιόν δίνει τη δυνατότητα στις άλλες αρμόδιες αρχές να ασκήσουν τον προπολογισμό, αλλά γίνεται εδώ λόγος και για συνεργασία των τριών οργάνων. Άρα, πρώτον, το 319 με βάση το παράγωγο δίκαιο και την πρακτική δεν λέει καθόλου ότι η Κομισιόν είναι η μόνη αρχή χρήση του προϋπολογισμού. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Μπορεί να είναι συζητήσιμα όλα αυτά, αλλά το παράγω δίκαιο, η πρακτική και το ίδιο το γράμμα του κειμένου δεν δείχνουν ότι η Κομισιόν είναι η μόνη αρχή χρήση του προϋπολογισμού. Και πάνω σε αυτή τη νομική και πρακτική βάση από το 2001 το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά έλεγχο και των δύο άλλων οργάνων. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί από νομικής πλευράς ως προηγούμενο, νομικό προηγούμενο. Διότι για να υπάρξει προηγούμενο για να θεωρηθεί κάτι ως ιωθός βασιζόμαστε και στην κυρίαρχη νομική άποψη. Ασαφές και αυτό, αλλά έτσι λένε. Εδώ και πολλά χρόνια όμως το Συμβούλιο αρνείται να συνεργαστεί και έχω εκπλαγεί βλέποντας σε ποιο βαθμό αρνείται το Συμβούλιο να συνεργαστεί, να δώσει έγγραφα Επανειλημμένος αρνείται. Μέχρι και σήμερα. Ακόμα που πρόκειται για μια άτυπη συζήτηση. Και με έκπληξη διαβάζω και από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου γιατί όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συζήτησή μας. Εάν το ελεγκτικό συνέδριο έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι όλα ρητά και σαφή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα και ότι άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δίκιο που λέει ότι παραγωνίζεται. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι η κατάσταση δεν είναι υγιής ως προς τη σωστή διαχείριση των δημοσίων πόρων ούτε σέβεται τον την αρχή του δημοκρατικού ελέγχου. Θα μιλήσω και για το πνεύμα και για το γράμμα των συνθήκων. Λοιπόν, η κυριότερη διαφωνία μου με τον προηγούμενο μιλητή είναι το θέμα της αφήνειας των συνθήκων. Εγώ δεν πιστεύω ως νομομαθής ότι μπορεί να υπάρχει τελείως καθαρό και ρητό κείμενο νομικό και αυτό ισχύει πόσο μάλλον για τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Βλέπετε πόσες φορές χρειάζεται να το ερμηνεύσει αυτό το δίκαιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένε περιπτώσεις, αλλά ποια είναι η λογική των συνθήκων. Είναι διπλή ω προς το θέμα μας. Δηλαδή, πρώτον, ότι αυξάνονται οι δικαιοδοσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενισχύονται, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ένα βιβλίο που είχα γράψει, έλεγα ότι το Κοινοβούλιο άρχισε από το τίποτα και κατέληξε να είναι σχεδόν τα πάντα εφόσον μεταξύ άλλων ελέγχει και τη χρήση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και για την θεσμική ισορροπία σας θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την το προσέχει πάντοτε αυτό το θέμα. Αρχικά το κοινοβούλιο δεν είχε παρά συμβουλευτικό ρόλο, λεγόταν συνέλευση, δεν εκλεγόταν άμεσα από τους λαούς και το δικαστήριο είχε υποχρεώσει, το θυμίζω αυτό, γιατί εκείνο ερμηνεύει τη συνθήκη, είχε υποχρεώσει το Συμβούλιο να συμβουλεύεται πάντα το Κοινοβούλιο όποτε κάποιο νομοθέτημα έχει σημαντικά αλλάξει. Επανθυμίζω ότι εκείνη την εποχή δεν είχε καμία δικαιοδοσία το Κοινοβούλιο. Άρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσέχει το θέμα αυτό του δημοκρατικού ελέγχου. Και η δεύτερη λογική είναι εκείνη της αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Η συνθήκη της Λισαβόνας είναι η πρώτη συνθήκη που αφιερώνει ολόκληρο τίτλο στο θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Και στον τίτλο αυτό δεν λέει ότι είναι ένας παράγοντας της δημοκρατίας και του δημοκρατικού ελέγχου και το Συμβούλιο. Δεν λέει ότι δεν είναι δημοκρατικό γιατί εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη αλλά δεν είναι εκείνο η κατεξοχήν δημοκρατική αρχή. Ποιες, ποια όργανα αναφέρει ο τίτλος αυτός της συνθήκης της Λισαβόνας στον τίτλο αυτό για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Το, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Τιούτο. Καταλήγουμε λοιπόν στην εξή διαπίστωση. Ότι θα μπορούσαν όλα αυτά να βελτιωθούν. Το θέμα όπως βλέπετε είναι λεπτό. Βλέπετε ήδη ότι υπάρχουν εδώ μεταξύ μας δύο ομομαθείς που δεν συμφωνούν. Δύο πιθανές λύσεις λοιπόν προσωπικές μου. Οι δικαστές ζητούν όλο και μεγαλύτερο σεβασμό των κοινοβουλευτικών δικαιοδοσιών. Σας ανέφερα μία προηγουμένως στην υποχρεωτική διαβούλευση αν αλλάξει νόμος και υπάρχει και μια άλλη, μια απόφαση του 2003 στην οποία είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Συμφωνία Κυρίων που αναφέρουν παρελθόν, του 83 με συγχωρείτε, όπου το δικαστήριο υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να διαταράσετε η θεσμική ισορροπία. Τι σημαίνει αυτό σε σχέση και με τη συμφωνία κυρίων που αναφέρει συχνά το Συμβούλιο. Η απόφαση του 83 και η συμφωνία του 70 συγκρινόμενες δείχνουν ότι το Συμβούλιο λέει ότι οι δικές του υποθέσεις είναι η χρήση του προπολογισμού του και μπορεί να φτάσει μέχρι και άρνηση υποβολής ε, των σχετικών εγγράφων στην αρχή την αρμόδια για τον έλεγχο του προπολογισμού. Αυτού του είδους η αντίληψη αντιβαίνει προς την αρχή της θεσμικής ισορροπίας. Αυτό σημαίνει η απόφαση του 83. Και μετά η συμφωνία κυρίων η συμφωνία εκείνη δεν είναι παράγωγο δίκαιο. Το δικαστήριο ποτέ δεν απεφάνθη επ' αυτής. Δεν είναι επισήμως δίκαιο δηλαδή. Και η επίκλησή της αντιβαίνει σε όλες τις εξελίξεις των τελευταίων 30 ετών ως προς την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. για να τα συνδέσουμε όλα αυτά με αυτά που είπαμε προηγουμένως, που είπαν και οι προηγούμενοι, το Συμβούλιο δεν συγκρίνεται με τον Bundesrat ή με τη Γερουσία. Γιατί συνήθως συγκρίνουμε ασύγκριτα πράγματα, ο καθένας αυτά που γνωρίζει, εντάξει φυσικό είναι, γιατί αυτά που οικοδομούνται εδώ είναι καινούρια πράγματα. Το Συμβούλιο πάντως επιμένω βασίζεται σε μία αρχή δυτής λειτουργίας. Η ερμηνεία που κάνει για τη Συμφωνία Κυρίων λέει ότι μπορεί να υπάρχει, πράγμα που είναι κακό, σύγχυση της φύσης των λειτουργιών το Συμβούλιο όταν αποφαίνεται δεν το κάνει ως νομοθέτης αλλά ως εκτελεστική αρχή. Γι' αυτό έχει δικαιοδοσία για την άσκηση, για τη χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτό είπα και πριν, δεν είναι μόνο η Κομισιόν, είναι και το Συμβούλιο που ασκούν τον προϋπολογισμό. Και το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να ανακατεύεται σε όλα αυτά το Κοινοβούλιο έχει κάποια βάση μεν, αλλά πρέπει να ξέρουμε καταρχήν τι είναι το Συμβούλιο. Είναι και νομοθέτης και εκτελεστική εξουσία. Άρα η επίκληση της Συμφωνίας Κυρίων του 70 αντιβαίνει και στην αρχή του δημοκρατικού ελέγχου και της διαφάνειας και στην πραγματικότητα της χρήσης του προϋπολογισμού. Τώρα, με βάση την απόφαση του 83 που ερμηνεύει τη συμφωνία του 70 θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε δύο περιπτώσεις αντίθεση Συμβουλίου Κοινοβουλίου το δικαστήριο έχει μιλήσει για θεσμική ισορροπία και συνεργασία των δύο οργάνων. Με βάση λοιπόν αυτή την ομολογία και την πράξη θα μπορούσε κανείς να φανταστεί μια προσφυγή. Δεν τη ζητάει κανείς βέβαια ούτε εγώ. Αλλά με βάση αυτή την επιχειρηματολογία για τις παρελθούσες αποφάσεις, για την ομολογία, για την θεσμική ισορροπία, για την ισορροπία των θεσμών νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει προσφυγή κατά του Συμβουλίου με βάση την ομολογία και των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων και αυτό είναι σημαντικό γιατί όπως είπα και πριν ο νέος τίτλος της Συνθήκης Λισαβόνας για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία αναφέρει και το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια και η πιο πρόσφατη νομολογία των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων όπως του Γαλλικού και της Καρλσρούης τι λίχνει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή πάντα η αρχή του δημοκρατικού ελέγχου Πάντοτε τονίζονται σε αυτές τις αποφάσεις ιδιαίτερα τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά αν υπήρχε μεγαλύτερο σεβασμός της ευρωπαϊκής δημοκρατίας σε ενωσιακό επίπεδο, τότε τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια θα πρόσεχαν όχι μόνο το θέμα του σεβασμού των δικαιοδοσιών των εθνικών κοινοβουλίων αλλά και του ευρωπαϊκού για να υπάρχει η συμπληρωματικότητα. Συμπέρασμα. Πρώτον, νομίζω ότι με βάση τις συνθήκες δεν ισχύει η επιχειρηματολογία του Συμβουλίου. Η Κομισιόν δεν είναι το μόνο όργανο που ασκεί, που κάνει χρήση του προϋπολογισμού. Και αυτό δεν αντιβαίνει στις συνθήκες. Το άρθρο 79 πουθενά δεν λέει ότι η Κομισιόν είναι το μόνο όργανο ή αρχή χρήσης του προϋπολογισμού. Δεύτερον, η ερμηνεία του Συμβουλίου είναι αντίθετη κατ' εμέ με την αρχή της θεσμικής ισορροπίας, με τη δημοκρατία και με την απέτηση για καλή διαχείριση, όπως λέει και το, και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και δεύτερο συμπέρασμα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των Εθνικών Συνταγματικών Δικαστηρίων, γιατί έτσι θα φανεί θα φανεί ότι οι συνθήκες πράγμα που συχνά το λέει και το δικαστήριο, οι συνθήκες λέω μπορεί να μην είναι τελείως σαφείς αλλά έχουν ερμηνευθεί επανειλημμένως με τρόπο αυτή τη φορά σαφή. Και εσείς είπατε κύριε συναδελφέ ότι και το Συμβούλιο είναι δημοκρατικό όργανο. Συμφωνώ, αλλά σκεφτείτε την απόφαση Μάθιους του 79, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβού καταδίκασε το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί δεν έκανε ευρωεκλογές στο Γιβραλτάρ. Τι μας λέει λοιπόν αυτό το δικαστήριο που δεν είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ότι δεν εκπροσωπήθηκε ολόκληρη η Ένωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει λοιπόν επαρκής έλεγχος είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το αποδείξουμε και να το χρησιμοποιήσουμε κατά του Συμβουλίου. Τρίτο συμπέρασμα να χρησιμοποιήσουμε την πρακτική, τη θεσμική πρακτική. Φυσικά το Συμβούλιο και αυτό το κάνει. Και αν φανούν δυσλειτουργίες στη χρήση του προϋπολογισμού, θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για να το αποδείξουμε. Τώρα επειδή περνάει η ώρα, θα ήθελα να πω κάτι και για την περίπτωση άρνησης απαλλαγής από το Κοινοβούλιο. Τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να είμαστε βέβαια εξαντλητικοί. Τέσσερις περιπτώσεις. Στα μέσα ενημέρωσης να αναφερθούν όλα αυτά. Συμμαχίες με την Κομισιόν προβουλευτικές δράσεις, προδικαστικές. Και τα εξηγώ. Στον τύπο θα μπορούσαμε να κάνουμε καμπάνιες, να δηλώσουμε, να ανακοινώσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος άρνησης της απαλλαγής λίγες μέρες πριν ληφθεί η απόφαση αυτή. Είτε με σύντομη ανακοίνωση είτε αυτό που προτιμώ με διάλογο πολλών ευρωβουλευτών όπου να ανακοινώνουν στην κοινή γνώμη ότι δεν θα δοθεί απαλλαγή. Η τρίτη υπόθεση δημοσίευση σε ειδικευμένα περιοδικά. Δεύτερη δυνατότητα. Συμμαχία ή αντιπαράθεση με την Κομισιόν. Συμμαχία ας πούμε με το επιχείρημα ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύουν το κοινό συμφέρον ενώ υπάρχει απ' την άλλη η αντίρρηση του Συμβουλίου. Αν τώρα η Κομισιόν δεν θέλει να κάνει τέτοια συμμαχία, τότε υπάρχει αντιπαράθεση. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως κυρία Σεντέρ, άρνηση απαλλαγή και προς την Κομισιόν. Θα μπορούσε να υπάρξει τέτοια αντιπαράθεση εάν η Κομισιόν δεν ενθαρρύνει το Συμβούλιο να υποβάλει τα έγγραφα και άρα δεν συνεργάζεται και, αυτό με, και αυτή με τη Δημοκρατία. Άρνηση απαλλαγής. Και τέλος, τρίτη, όχι μάλλον προτελευταία περίπτωση, προδικαστικό βούλευμα. Δηλαδή, να γνωστοποιήσουμε στο Συμβούλιο ότι χρειαζόμαστε έγγραφα και αν δεν μας τα δώσετε δεν θα δώσουμε απαλλαγή. Και τέλος προσφυγή κατά του Συμβουλίου με τα επιχειρήματα που ανέφερα, έλλειψη δημοκρατικότητας, ε, θεσμική συνεργασίας κλπ. Και το επιχείρημα ότι η Συμφωνία Κυρίων του 70 δεν έχει νομικό χαρακτήρα. Μπορεί να μακρηγόρησα, αλλά αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαλτιέλα. Και τώρα δίνω το λόγο στον επόμενο ειδικό, τον κύριο Καρλίνο Εντπένερ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κυρία Γιάλα Σέντερ, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω ε, για την πρόσκλησή μου σε αυτό ε, το σεμινάριο και με μεγάλη χαρά θα σας υποστηρίξω στην προσπάθειά σας. Το ερώτημα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αρνηθεί την απαλλαγή του Συμβουλίου. Εγώ πιστεύω ότι ναι και θα σας εξηγήσω γιατί και γι' αυτό θα προχωρήσω με σε τρεις ε, βήματα. Καταρχήν ή ε, στο κείμενο της συνθήκης και του δημοσιονομικού κανονισμού που διαβάζω και ερμηνεύω από άλλη οπτική γωνία. Θα παραθέσω Διάφορε διάφορες ευρωπαϊκές αρχές που δίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να αποφασίσει για την απαλλαγή του Συμβουλίου και τρίτον σχετικά με τις επιπτώσεις και τα δικαιώματα πληροφόρησης του Κοινοβουλίου. Το θέμα ρυθμίζεται στο άρθρο 319 της συνθήκης και προβλέπεται απλώς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απαλλάξει ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για ολόκληρο τον προϋπολογισμό χωρίς να υπάρχει ρύθμιση ε, για το Συμβούλιο και δεν ρυθμίζεται εάν απαλλάσσεται από αυτήν την απαλλαγή το Συμβούλιο. Αλλά δεν λέγεται ότι η συνομοθεσία ότι το Κοινοβούλιο απαλλάσσει μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και όπως είπε ο κύριος Ρώση ενδεχομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα κλειστό σύστημα που, όπου ε, μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαλλάσσεται. Ενδέχεται όμως να μπορούν να ληφθούν και ε, διαφορετικές και χωριστές ε, απαλλαγές για τα, διάφορα, τα διάφορα θεσμικά όργανα. Ως εκ τούτου βλέπουμε ότι υπάρχει μόνο μία απαλλαγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύμφωνα με το άρθρο 317 παράγραφος 1 της συνθήκης που αναφέρθηκε επανειλημμένος λέγεται ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να... Α, να απαλλάξει όλα τα θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο. Στο παρελθόν υπήρχε μία διαφορά στην ερμηνεία. Τώρα όμως πρέπει να παραθέσει κανείς τα ιστορικά στοιχεία. Πρέπει να δούμε ότι εάν πρέπει να αλλάξει το ενδεχομένως η νομοθεσία και σε αυτό προσφέρεται το πρωτογενέ διεθνές και το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο όπως και ο καθηγητής ε, ε, Ρώση πιστεύω ότι υπάρχει μία διαφορετική μια διαφορά μεταξύ των δύο ερμηνεών της νομοθεσίας μέχρι όμως ενός βαθμού αυτό μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να εξαλείπτει την, ε, το όριο μεταξύ ερμηνείας και νομοθεσίας δηλαδή ε, η ερμηνεία μπορεί να αλλάξει αλλά πρέπει να ενεργεί κανείς μέσα στα όρια της διατύπωσης και αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το τωρινό θέμα διότι ε, ο κανόνας βάσει του οποίου ρυθμίζεται η απαλλαγή ανέρχεται στο 1977 και αυτό δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Αντιθέτως όμως οι συνθήκες έχουν αλλάξει πολύ και ο χαρακτήρας του Συμβουλίου έχει αλλάξει ο οποίος το οποίο αναλαμβάνει όλο και περισσότερο εκτελεστικά καθήκοντα και αναφέρομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο συζητά τον κοινό προπολογισμό μαζί σας είναι πιο σημαντικό και αντικαθιστά την κυβέρνηση και τις λειτουργίες της κυβέρνησης. Επίσης όσον αφορά την οικονομική πολιτική έχει βασικές εκτελεστικές οργανότητες. Αυτές λοιπόν οι ιδιότητες είναι παράγοντες για να απαντήσει κανείς το ερώτημα εάν το Κοινοβούλιο ε, ε, ε, είναι εξουσιοδοτημένο να απαλλάξει το Συμβούλιο. Διότι από το 1977 οι θεσμοί δεν άλλαξαν αλλά η θεσμική δομή άλλαξε σε τρομερά και όπως ήδη σας είπα και η διατύπωση είναι αμφίσιμη. Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι επιτρέπεται μόνο μία μοναδική απαλλαγή ή ότι πρέπει να υπάρξουν διαφορετικές απαλλαγές. Ιστορικά ε, είχε αποφασιστεί ότι υπάρχει μόνο μία απαλλαγή, ε, δεν είναι όμως η ουσιαστική ερμηνεία τώρα και πιστεύω ότι το άρθρο 300 δεν είναι προφανές και μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά. Για να αντεπεξέλθει κανείς σε αυτήν την αμφισημία πρέπει να βασιστεί στις ευρωπαϊκές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και καταρχήν ε, την δημοκρατική ευθύνη που είναι ένα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας για δημοσιονομική ε, διαδικασία αυτό σημαίνει ότι η νομιμοποίηση γίνεται μετά από έλεγχο εκ των υστέρων και αυτό μπορεί να υποβληθεί στον έλεγχο της κοινή γνώμης και να εξυπηρετήσει κατά αυτόν τον τρόπο το δημόσιο διάλογο και την διαφάνεια. Πώς καταρτίστηκε αυτή η δημοκρατική ευθύνη αν ακολουθήσουμε το σκεπτικό του καθηγητή Ρώση ότι δηλαδή δεν πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παλάσει το Συμβούλιο τότε ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ε, υπάρχει δύο στοιχεία το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ουσιαστικά νομιμοποιείται μόνο δια του ελέγχου των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, των εθνικών κυβερνήσεων από τα εθνικά κοινοβούλια ενώ είναι διαφορετική η μορφή του κοινοβουλίου και η συμμετοχή των ευρωπαϊκών ε, των εθνικών κοινοβουλίων ε, αναφέρεται μόνο στην νομοθετική διαδικασία και ο προϋπολογισμός της διαχείρισης του Συμβουλίου μπορεί μόνο να ελεγχθεί σε επίπεδο Συμβουλίου. Γι' αυτό και ο έλεγχος των εθνικών κοινοβουλίων δεν αποδίδει στην περίπτωση αυτή και η νομιμοποίηση μπορεί να γίνει μέσω της του δευτέρου πυλώνα δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι ε, αυτό είναι το θεσμικό όργανο που έχει την κυριότητα της ε, διαδικασίας απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 310 ο δεύτερος πυλώνας εκπροσωπείται επαρκώς μόνο εάν ο έλεγχος εκ των υστέρων διεξάγεται από το Κοινοβούλιο. Παραδείγματο χάρη, αν το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου και στη συνέχεια ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία ε, η οποία να προσφέρει μία δημοκρατική νομιμοποίηση και αυτή τη στιγμή ο έλεγχος του Συμβουλίου γίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και δεν ε, νομιμοποιείται εξ δημοκρατικά. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικός δημοσιονομικός έλεγχος του Συμβουλίου και δημιουργούνται φοβερά δημοκρατικά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με δύο τρόπους. Ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ελέγχει τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου ή να τον ελέγχει κατευθείαν το Κοινοβούλιο. Εγώ προτιμώ τη δεύτερη λύση διότι πιστεύω ότι η πρώτη δυνατότητα μπορεί να δημιουργήσει ασάφειες και έτσι ε, είναι δικαίωμα του Κοινοβουλίου να απαλλάσσει το Συμβούλιο πράγμα το οποίο προσφέρει σημαντικά δημοκρατικά προσόντα. Λέγεται επίσης στις συνθήκες ότι τα θεσμικά όργανα μπορούν να ρυθμίσουν ρυθμίσουν αυτόνομα τις εσωτερικές τους ε, ε, υποθέσεις και αυτό μπορεί ε, να θεωρηθεί σαν να ισχύει για τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου για έξοδα κτηρίων και προσωπικού. Ε, υπάρχει όμως σκόπιμό της να καθοριστούν τα ίδια ίδια έξοδα από το Συμβούλιο χωρίς όμως αυτό να καλύπτει την νομιμότητα των δαπανών και σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 5 της συνθήκης ε, τα θέματα αυτά ε, και τα έξοδα αυτά πλήττουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής της στο σύνολό της γι' αυτό και δεν μπορεί να περιοριστεί κανείς στον ε, έλεγχο της Επιτροπής υπάρχουν επίσης οι παραβιάσεις των αρχών οικονομίας αποδοτικότητος και αποτελεσματικότητος δηλαδή ο έλεγχος του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι πολύ εκτενής πράγμα το οποίο δεν ε, ε, αποκλείει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να απαλλάξει το Συμβούλιο αλλά αυτό πρέπει να γίνεται στα πλαίσια μιας θεσμικής ισορροπίας και με ε, έλεγχο της νομιμότητος πρέπει ε, η διαδικασία αυτή να βασίζεται στο πρωτογενές δίκαιο και εφόσον το Συμβούλιο είναι συνομοθέτης δεν μπορεί ε, να αποκλείεται από κάθε έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι αυτό θα έφερνε θέτε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του Συμβουλίου. Θα πρέπει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να θεωρηθούν ισότιμοι νομοθέτες οι οποίοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και αυτός ίσως ήταν ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο δεν μπορούσε ιστορικά να ελέγξει άμεσα το Συμβούλιο. Αυτή είναι μια σημαντική αντίρρηση, αλλά υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα που δεν αφαιρούν από το Κοινοβούλιο το δικαίωμα να ελέγξει το Συμβούλιο. Διότι ενώ σε άλλα σημεία των συνθήκων δεν ρυθμίζεται ε, η το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ελέγξει το Συμβούλιο, η ανεξαρτησία του Συμβουλίου η στη δημοσιονομική διαδικασία σαφώς περιορίζεται και είναι αδιαφυσβήτητο ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου μπορεί να ελεγχθεί από το Κοινοβούλιο. Το ερώτημα είναι όμως αν αυτό μπορεί να γίνει μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι επιπτώσεις ε, ε, του δικαιώματος αυτός του Κοινοβουλίου επί της θέσεως του Συμβουλίου είναι πολύ πιο περιορισμένες και ε, αυτό δεν αφαιρεί ε, από το Συμβούλιο παρά μόνο ένα μικρό κλάσμα της αυτονομίας τους στον τομέα του ελέγχου του προπολογισμού. Και εδώ διαφωνώ με τον καθηγητή Ρώση διότι νομίζω ότι πρέπει να προβλέπεται ένα ουσιαστικός έλεγχος του προϋπολογισμού για να μπορεί το Συμβούλιο να κατέχει ε, την, ε, τις δυνατότητές του και να υπάρχει θεσμική ισορροπία. Η αρχή της θεσμικής ισορροπίας είναι πολύ σαφή στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν ε, διευκρινίζεται στην νομολογία και ο δημοσιονομικός έλεγχος ε, δεν μπορεί να γίνεται μόνο από την μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει ισορροπία. Υπάρχει και το θέμα της ε, δημοκρατικής, ε, του δημοκρατικού ελέγχου και δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύει την δημοκρατία ως απλούστατα ε, έκφραση της ε, της θεσμικής ισορροπίας αντιθέτως η δημοκρατική ευθύνη είναι δικαίωμα του Κοινοβουλίου και γι' αυτό πρέπει να μπορεί ε, να νομιμοποιείται εκ των υστέρων ε, δημοσιονομικός έλεγχος του Συμβουλίου. Το δικαίωμα ελόγξεως του προϋπολογισμού η ελέγχου του προϋπολογισμού ε, είναι ένα ισχύον καθήκον και αιτιολογείται και νομιμοποιείται. Αυτό το οποίο ε, λοιπόν πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι θα εμεινεύσουμε την ισορροπία των θεσμικών οργάνων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην τη διαταράξουμε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ε, το δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου πρέπει να περιοριστεί στα εκτελεστικά καθήκοντα οπότε δεν δημιουργούνται προβλήματα και σαν συνδετικός κρίκος ε, παρατίθεται το άρθρο 77 του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το οποίο ο έλεγχος του Συμβουλίου ε, για την δραστηριότητά του θεωρείται σαν έλεγχος ενός εκτελεστικού οργάνου. Δεν πρέπει όμως να μειώσουμε τις, ε, τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου για να ελέγξει κανείς τα έξοδα για προσωπικό και τα κτίρια δεν χρειάζεται ε, να διευκρινίσει κανείς αν το κονδύλι αυτό είναι εκτελεστικό ή νομοθετικό και ε, δεν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού των δύο κατηθικόντων. Θέλω να αναφερθώ τώρα στο άλλο θέμα που είναι το δικαίωμα Πληροφόρηση ε, και ε, στην διαδικασία. Η κυρία Σαλτιέλ και ο κύριος Ρώση ήδη έχουν παρουσιάσει ορισμένα επιχειρήματα και ως εκ τούτου θεωρώ ότι πρέπει κανείς να καλύψει το τμήμα του προϋπολογισμού μέσα σε αυτόν τον έλεγχο που δεν εκτελεί άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λοιπόν ε, καθήκον του Συμβουλίου να διαθέτει τις πληροφορίες ενδεχομένως μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, υπάρχει από το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο αυτή η δυνατότητα για το Κοινοβούλιο. Γενικώ μέχρι στιγμής ε, δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αρκεί ε, να καλύψει την υποχρέωσή του το Συμβούλιο με προφορικές απαντήσεις και με παρουσία στην Επιτροπή. Πρέπει ε, ε, να μπορούσε κανείς να βασίσει ε, το δικαίωμα του Κοινοβούλιο και βλέπουμε εδώ μία ανακοίνωση του Συμβουλίου το 1977 όπου το Συμβούλιο υποχρεούται να απαντήσει εκτενώς σε προφορικά και γραπτές ερωτήσεις όπως είπε και ο κύριος Ρώση. Έτσι ε, το Συμβούλιο μπορεί να εκτελέσει ε, τις, ε, τα καθήκοντά του για παρουσίαση προτάσεων εξόδων αλλά συγχρόνως πρέπει να προσφέρει και τις πληροφορίες. Πέραν αυτού όλα αυτά έχουν ε, παρουσιαστεί από την κυρία Σαλτιέλ οπότε θα είμαι πολύ σύντομο Το παράγωγο δίκαιο υποχρεώνει όλα τα θεσμικά όργανα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν τα στοιχεία. Η απόφαση όμως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, περί περιορίζει ε, την ε, διαχείριση αυτών των πληροφοριών. Αυτή τη στιγμή ε, δεν υπάρχει μία πράξη του Συμβουλίου που να το δεσμεύει αλλά το Κοινοβούλιο δικαιούται να έχει επιπρόσθετες πληροφορίες εφόσον τις χρειάζεται και έχει εκτενέστερο δικαίωμα πληροφόρησης από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 319 και σύμφωνα με ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όντως το Κοινοβούλιο μπορεί να ε, ελέγξει και να απαλλάξει το Ευρωπαϊκό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και εσάς και τους δύο προλαλήσαντες. Είχαμε σκεφτεί ότι αυτή τη στιγμή θα μπορέσουν να υπάρξουν ερωτήσεις και στη συνέχεια να επέμβει η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υπάρξει ένας δεύτερος γύρος γενικής συζήτησης. Τώρα λοιπόν θέλω να σας πω κύριε Ρώση ότι η γραμματεία έχει καταρτήσει ε, μία σελίδα για τον δημοσιονομικό κανονισμό και ε, εάν δεν βρίσκεται την ιστοσελίδα μας επειδή και εμείς ενδιαφερόμαστε να ε, παρέχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε και να μας επισημάνετε εάν υπάρξει κάποια έλλειψη. Τώρα λοιπόν έχω σαν πρώτο μιλητή τον Σόρεν Σέντεγκαρτ. Ευχαριστώ για αυτές τις τρεις ενδιαφέρουσες ε, ε, τοποθετήσεις. Ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικές. Ποτέ δεν ετέθη το ζήτημα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αν θα πρέπει να λαμβάνουμε ή όχι κατευθείαν τις πληροφορίες από το Συμβούλιο. Δεν είναι αυτό το οποίο αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Απλώς αυτό το οποίο μας απασχολεί εξ ονόματος των Ευρωπαίων πολιτών είναι να ξέρουμε πώς χρησιμοποιούνται τα λεφτά. Από αυτά που άκουσα εγώ υποθέτω ότι το Κοινοβούλιο έχει αυτό το δικαίωμα. Τώρα πρέπει να δούμε αν οι επιπτώσεις αυτού του, αυτού του γεγονότος ε, οδηγεί στο δικαίωμα, στο αναγνωρισμένο δικαίωμα του Κοινοβουλίου για τη χορήγηση της απαλλαγής και για μένα αυτό αποτελεί μια αποφασιστική διευκρίνηση. Θέλω να ρωτήσω, εάν το Κοινοβούλιο αποφάσισε να παρουσιάσει, να καταθέσει μία προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αυτό λόγω μη παρουσίαση εγγράφων που εμεί ζητήσαμε από το Συμβούλιο μέσα στη διαδικασία απαλλαγή και το Συμβούλιο δεν μα τα έδωσε. Οι ομιλητέ μα λένε ότι Λέτε μάλλον ότι είναι ενδιαφέρον να καταθέσουμε εμείς μία τέτοια προσφυγή και πιστεύετε ότι θα είχε μια καλή απήχηση και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και όλες την υπόθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντρέασεν ζητά το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, το θέμα είναι μάλλον πολιτικό παρά τεχνικό και ε, δείχνει η διαμάχη των δύο οργάνων την κρίση που υφίσταται ολόκληρη η Ένωση. Μιλήσαμε για το ποιος είναι υπεύθυνος λέει. Ποιος είναι όμως υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό, για την απαλλαγή, για την προάσπιση των συμφερόντων των φορολογουμένων. Από ό,τι άκουσα η συνθήκη είναι σαφής κατά το εξής η Κομισιόν είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Βέβαια πρέπει να ζητήσει πληροφορίες και από τα άλλα όργανα, αλλά η ευθύνη είναι της Κομισιόν. Πρέπει να δούμε το θέμα στην ουσία του. Εγώ θεωρώ ότι η λύση είναι να ζητούμε πληροφόρηση από την Κομισιόν, όπως κάνουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Τι φρονούν οι ομιλητές γι' αυτό. Η λύση είναι απλή. Η Κομισιόν είναι το όργανο στο οποίο πρέπει να απευθυνθούμε. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, τρεις εμπειρογνώμονες γιατί άλλος ε, υπέρ ή άλλος ε, κατά των θέσεών μας βοήθησαν ε, να διαπιστώσουμε ποια είναι αυτά τα προβλήματα. Εγώ δεν συμφωνώ με την κυρία Αντριάζεν ότι θα πρέπει να αμφισβητήσουμε όλο το δόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το 1,59% που ξοδεύει το Συμβούλιο επί του συνόλου του προϋπολογισμού. Θέλω να ρωτήσω τώρα στον κύριο Ρώση. που διατύπωσε την ε, που έκανε και την ε, ε, πιο θα έλεγα προκλητική πρόκληση θα έλεγα ότι τον, τον πλήρωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου για να μας την κάνει Να το ρωτήσω. Αυτό το οποίο δεν είναι γραμμένο σαφέ, σαφώς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το προσδιορίσουμε και να καταφέρουμε να το εγγράψουμε κάπου και να το καταγράψουμε. Στο άρθρο όμως, 19, ε, μιλάμε ε, για, τις, ε, για τους ελεγχόμενους οργανισμούς σε αυτό το άρθρο που λέει ότι η Κομισιόν είναι η μόνη υπεύθυνη κτλ. Υπάρχει ένα, μία παράγραφος που λέει η απάντηση των ελεγχομένων ε, θεσμικών οργάνων. Έτσι το έχω εγώ στα ισπανικά. Δεν ξέρω στα γερμανικά το επίθετο και αυτό θα είναι στον πληθυντικό. Ελεγχόμενοι οργανισμοί. Λοιπόν, αυτό ελέγχεται σύμφωνα το Συμβούλιο και μετά το ελεγκτικό συνέδριο του κάνει τον έλεγχο. Μετά υπάρχει και ένα βασικό στοιχείο που λέει ότι κάποια ευθύνη έχει και το Συμβούλιο. Και εμάς ναι μεν δεν μας απαντάει το Συμβούλιο, αλλά στο ελεγκτικό συνέδριο βεβαίως και απαντάει. Είναι υπεύθυνο τουλάχιστον έναντι του ελεγκτικού συνεδρίου. Διότι κάτι θα έπρεπε ως προς τον έλεγχο να τίθεται. Υπάρχουν όμως και άλλα άρθρα, ας πούμε το άρθρο 116 όπου λέει ότι θα πρέπει να ελέγχονται ξεχωριστά τα τρία όργανα, όχι μόνο για όταν ξοδεύουν αλλά και όταν ε, ελέγχονται. Μιλάει επίσης και για διοικητική αυτονομία. Το άρθρο 50 λέει ότι εφόσον υπάρχει διοικητική αυτονομία, αυτό προστατεύει το Συμβούλιο. Και το άρθρο 324 της Συνθήκης που λέει ότι υπάρχει υποχρέωση των προέδρων των θεσμικών οργάνων να ή χάνουν μίας προσέγγισης μεταξύ τους να ενώνονται για να μπορούν να διευκολύνουν τον δημοσιονομικό έλεγχο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η υποχρέωση για την διευκόλυνση του ελέγχου. Σας ρωτώ λοιπόν, αυτά τα στοιχεία τα λάβατε υπόψη σας όταν είπατε ότι η Κομισιόν είναι υπεύθυνη και όλοι οι υπόλοιποι όχι. Δεν λέει πουθενά ότι το Συμβούλιο δεν είναι υπεύθυνο. Οπότε αυτό είναι ένα περιθώριο λιγμών που μπορεί να αξιοποιήσει το Κοινοβούλιο. Στην κυρία Σαλτιέλ ε, μας άνοιξε πολλές ε, δυνατότητες και για το θέμα του δικαστηρίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τι βαρύτητα έχει αυτή η κουτί με αυτό το έθιμο ε, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό λοιπόν το έθιμο, αυτό το εθιμικό δίκαιο, τι αξία έχει τι μπορεί να κάνει. Έχει κάποια αξία. Και στον ε, κύριο Αντ Τι νομοθετική αξία. Ποια είναι η νομική βαρύτητα της δήλωσης του Συμβουλίου ότι πρέπει να παρέχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες αυτό μέσα στην παλιά Συμφωνία Κυρίων. Υπάρχει μια νομική βαρύτητα από αυτού. Ο κύριος Μέλτερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και τις βρήκα πολύ ψηλής ποιότητας. Επειδή εδώ εκφράστηκαν δύο απόψεις κατά, εδώ τα όργανα είναι δύο κατά ενός, χωρίς να είμαι δικηγόρος πρέπει να πω ότι ένα είναι το κοινό σημείο των εισηγήσεων ότι το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να πληροφορεί, να μας δίνει τα στοιχεία που ζητάμε. Τα υπόλοιπα είναι θεωρητικά και ακαδημαϊκά. Το γεγονός είναι ότι το Συμβούλιο ακόμη και σήμερα αρνείται να παραστεί. δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει καλύτερα την αλαζονία του. Υπάρχει ένα όργανο που περιφρονεί το Κοινοβούλιο και τις δημοκρατικές του δικαιοδοσίες. αυτό αποκλειόταν να συμβεί σε κάποιο κράτος μέλος. Βρισκόμαστε όμως σε αδιέξοδο και η καθηγήτρια Σαλτιέλ νομίζω μας έκανε ορισμένες χρήσιμες συστάσεις, θα μπορούσαν και οι άλλοι δύο να μας κάνουν καμία πρόταση. Τι θεωρούν ότι πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο, ποιος θα ήταν ο ευκολότερος τρόπος θα ήταν η προσφυγή στο δικαστήριο. Γιατί αφότου εκφραστεί το δικαστήριο λύγει το πρόβλημα. Αντί κάθε χρόνο να συζητάμε τα ίδια. Συμφωνούν λοιπόν οι ομιλητές ότι ο μόνος τρόπος είναι να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Ευχαριστώ. Και τέλος ο κύριος Γκάιερ και η κυρία Γκρέσλε. Ναι. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ε, συγχαρώ τους ε, εμπειρογνώμονες άκουσα δύο ομιλίες στην μητρική μου γλώσσα και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την ασυνήθιστη εργασία τους ομιλητές με ενδιέφεραν και οι τρεις ομιλίες και ε, το μόνο σημείο που υπάρχει ομοφορία μεταξύ των τριών ομιλητών είναι αυτό στο οποίο πρέπει να βασιστούμε διότι και οι τρεις είπαν ότι υπάρχει μία υποχρέωση ενημέρωσης και ε, συμφωνώ με τον Σερεν ο οποίος λέγει ε, μέσω ποιας οδού θα εξασφαλίσουμε αυτή την πληροφόρηση μέσω της γραμματείας του Συμβουλίου ή ε, θα ζητήσουμε από την υπεύθυνη ε, από την ε, υπεύθυνη για την εκτέλεση, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία. Και ε, τελικά το ερώτημα είναι, το Συμβούλιο είναι υπόλογος δια της μίας ή της άλλης νομικής οδού ή όχι. Και πιστεύω ότι η συνθήκη είναι σαφέστατη και ε, εκεί συμφωνώ με τον καθηγητή Ρώση αλλά βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δυναμική ενότητα ως εκ τούτου η συνθήκη και φαντάζομαι ότι αυτό είναι το σημείο κινήσεως για τον νομικό δεν μπορεί να απαντήσει ικανοποιητικά σε όλα τα ερωτήματα, το είπες και εσύ. Είναι σωστό. Ε, πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είτε διευκρινίζουν είτε ε, ε, προβαίνουν σε ε, πιο λεπτομερείς διευκρινήσεις και εκεί που χρειαζόμαστε εμείς διευκρινήσεις τότε θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και γι' αυτό το θέμα της απαλλαγής του Συμβουλίου είναι τέτοιο ώστε πρέπει να ακολουθήσουμε την οδό μέσω της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και ε, θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να αντεπεξέλθουμε και να μην εμπλακούμε σε αυτό το αδιέξοδο. Βάσει όμως της αρχής της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας πρέπει και το Συμβούλιο να συμπράξει. Και ενώ το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή μας λέγουν είναι υποχρεωμένοι έναντί μας ε, οπότε ε, όσο δεν αντιδρούν δεν χρειάζεται να προσφέρουμε στοιχεία και πρέπει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Εάν λοιπόν ε, βάσει βάση της ε, την οποία κάποια μέρα ελπίζω να έχουμε. Ε, δεν συμφωνούμε με τις θέσεις που έλαβε ε, το Συμβούλιο, δεν θα το απαλλάσσουμε. Πώς εσείς ε, αξιολογείται τις αναγκαίες επιπτώσεις της μη απαλλαγής. Μέχρι στιγμής ιστορικά δεν υπάρχει ε, κάποια, κάποιο πρόβλημα. Έχουμε ένα προηγούμενο όταν ε, το 89 απειλήσαμε να μην απαλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρετήθηκε. Το ερώτημα είναι όμως πώς θα προχωρήσουμε και αν δεν απαλλάξουμε το Συμβούλιο πότε, πώς θα λειτουργήσει ε, το διαθεσμικό πλαίσιο στη συνέχεια. Η κυρία Γκρέσλε, το Συμβούλιο δεν χρειάστηκε να παραστεί, τα ξέρει όλα αλλά ε, θέλω να κάνω ορισμένε ερωτήσει στον καθηγητή Ρώση. Αυτό το οποίο εσείς παρουσιάστε σαν θέση είναι η θέση και του Συμβουλίου. Έχω ασχοληθεί με, σαν εισηγήτρια της Επιτροπής προεπολογισμού ώρες με το θέμα αυτό και ε, τα άρθρα που αναφέρονται στην απαλλαγή δεν έχουν αλλάξει εδώ και χρόνια γιατί δεν έχουμε ποτέ συμφωνήσει. Βεβαίως ε, δεν μιλήσατε για το άρθρο άρθρο της συνθήκης που αναφέρεται στην διοικητική αυτονομία του θεσμικού οργάνου και εδώ υπάρχει αντίφαση μεταξύ του 319 ε, και του άρθρου 353 που πραγματεύεται αυτό το θέμα και έχουμε προσπαθήσει να ε, συνδυάσουμε αυτά τα δύο άρθρα και να πούμε ότι υπάρχουν θεσμικά όργανα και ε, τα θεσμικά όργανα αυτά μας ε, υποβάλλουν τα έγγραφα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην απαλλαγή. Τώρα όμως βλέπουμε ότι το σχετικό άρθρο του ε, Τη συνθήκη λέει ότι ε, ε, η Επιτροπή έπρεπε να απαλλαγεί διότι το 1970 είχε η Επιτροπή όλους τους λογαριασμούς και όταν άλλαξε αυτή η λογιστική δεν άλλαξε η συνθήκη και ε, υπάρχουν πολιτικοί και νομικοί σε όλες αυτές τις επιτροπές και ε, συζητούν για θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με το δημοσιονομικό κανονισμό και οι νομικοί του Συμβουλίου ποτέ δεν αναφέρθηκαν σε όλο αυτό το θέμα. Δηλαδή γιατί δεν έπρεπε να ακολουθήσουν τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμέσου των ετών σε ένα βασικό θέμα του ε, κοινοβουλευτικού δικαιώματος που είναι το δικαίωμα απαλλαγής ε, υπάρχει σαν καθήκον του, Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου ε, η απαλλαγή στη συνθήκη αλλά ε, δεν μας δίδεται μέσα στη συνθήκη αυτή η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το καθήκον μας. Πώς λοιπόν θα συνδυάσουμε το 319 με το 353 μπορούμε ίσως να πούμε ότι θα γίνει μια συνολική ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι όλοι και μετά θα απαλλάξουμε κάθε ε, θεσμικό όργανο χωριστά. Υπάρχει ένας τεράστιος οργανισμός και αν πρέπει ο κάθε ένας, κάθε υποδιέρηση να απαλλάστε χωριστά. Δεν θα αλλάξουμε πολλά γιατί θα κάνουμε μία επιπρόσθεση απαλλαγή ε, εάν ε, εμεί απαλλάσσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη και την ημέρα που θα αρνηθούμε αυτή την απαλλαγή θα δείτε τι έχει να γίνει. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε διότι για να μειώσουμε την γραφειοκρατία και ε, να απλοποιήσουμε τη διαδικασία δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις. Είναι μια πολύ βαριά γραφειοκρατική διαδικασία και τι θα γινόταν αν έπρεπε να διαλύσουμε όλα τα λογιστήρια των οργανισμών και να τα φορτώσουμε όλα ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα χρειαζόταν 5.000 νέους συνεργάτες και απλούστατα θα περιπλέκαμε το θέμα. Ίσως νομικά θα ήταν πιο σαφές ε, το ε, πλαίσιο αλλά νομίζω ότι κατά η κατάσταση ίσως είναι ε, τρομακτική και τι να κάνουμε όμως ε, είμαστε ένας μεγάλος οργανισμός. Είπατε ότι πρέπει να γίνεται και έλεγχος νομιμότητος. Αυτή τόσο έλεγχος νομιμότητος ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι ανοησία και ε, παραποιείται. Μπορεί δηλαδή να χρηματοδοτήσει κανείς οποιαδήποτε ανοησία και όλα πάνε, πάνε θαυμάσια και τρέχουν ρολόι. Αυτό εννοείται ή εννοείται μία ε, ε, νομιμοποίηση και αναλογικότητα που είναι αρχές που δεν αρέσουν στους νομικούς δεν επαρκεί όμως να πούμε ότι coché και «Ζεκοσέλα του δικός». Δηλαδή ε, σημειώνω ότι έχω σημειώσει κάθε ε, τετραγωνάκι. Ε, εάν δηλαδή έχουμε σημειώσει όλες, όλα τα τετραγωνάκια πάνε όλα καλά, μέχρι στιγμής δεν ήξερα ότι ε, το να σημειώνει κανείς τετραγωνάκια είναι μέρος της ε, διαδικασίας απαλλαγής του υπροπολογισμού ή ότι πρέπει να εμπλακούν και τα ζώα αλλά ε, δεν ήθελα εδώ να πω κάτι ιδιαίτερο απλούστατα να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα και τώρα θα ήθελα να ακολουθήσουμε την αντίθετη σειρά η ώρα περνά. Θα ήθελα λοιπόν ο καθένας να μην ξεπεράσει 5 έως 7 λεπτά για να απαντήσει στα βασικά ερωτήματα κατά τρόπον ώστε να ακούσουμε στη συνέχεια και την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος και θα μπορέσω να συνοψίσω διάφορες ερωτήσεις. Καταρχήν, πολλοί αναφέρθηκαν στο δικαίωμα πληροφόρησης. Ο κύριος Ζόντερ Λόκεργκαρτ, Μέλλερ και Γκάιερ. Εάν κοιτάξουμε τη συνθήκη υπάρχουν δύο διαφορετικά δικαιώματα πληροφόρησης από το 3.19.10 για συγκεκριμένα έγγραφα και 3.19 παράγραφος 2 που καλύπτει τα πάντα. Σύμφωνα με το 3.19.1 αυτό που μας ενδιαφέρει, σύμφωνα με τη συνθήκη και το διοσιονομικό κανονισμό, η ε, υπόχρεη για πληροφόρηση είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά φαντάζομαι ότι θα μας πούν ε, και οι άλλοι συμμετέχοντες ότι ε, για να υπάρχει μία δίκαιη και πιστή συνεργασία πρέπει ε, να εμπλακούν και τα άλλα θεσμικά όργανα. Επίσης όσον αφορά για την επιτυχία κειμένων που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πιστεύω ότι ε, όλα, τα θεσμικά όργανα μπορούν να αποδείξουν ότι έχει ρυθμιστεί το δικαίωμα πληροφόρησης και αυτό σύμφωνα με το πνεύμα των τριών εισηγητών Λοιπόν στη συζήτηση. Υπάρχει λοιπόν μία ε, ε, σύσταση να ζητήσει κανείς ε, στο και ένδικα τις πληροφορίες και μπορεί να τις επιτύχει. Η δεύτερη ερώτηση του κυρίου Γκάιερ, πώς, ποια θα ήταν η η ε, επίπτωση για το Συμβούλιο εάν αρνεί το κανείς την απαλλαγή. Δεν πρόκειται για πρόταση μορφή, αλλά στο άρθρο 3 της συνθήκης λέγεται ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να αναλάβουν τις σκόπιμες πράξεις. Αυτό αναφέρεται στο πρωτογενές δίκαιο μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο παράγωγο δίκαιο σε όλα τα θεσμικά Δηλαδή, ε, όργανα τα οποία πρέπει να αναλάβουν μέτρα και φαντάζομαι ότι και νομικά μπορεί κανείς να προσφύγει κατά του δικαιώματος αυτού. Βέβαια η σκοπιμότητα είναι ε, κάτι στο οποίο ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα δώσει την ευρύτερη δυνατή διεκριτική ευχέρεια στα θεσμικά όργανα και υπάρχουν διάφορες πολιτικές ε, λύσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί αλλά ενδέχεται εις ε, την επόμενη διαπραγμάτευση να χρησιμοποιήσει κανείς ε, την απαλλαγή για να επιτύχει υποχωρήσεις. Στην ερώτηση του, της κυρίας Αγιάλα Σέντερς για το, τη δήλωση του Συμβουλίου του 70 αναφέρεται στο γενικό δικαίωμα πληροφόρησης του Κοινοβουλίου όχι μόνο σε δημοσιονομικά θέματα αλλά και γενικότερα όλα τα δικαιώματα δηλαδή θα το ψάξω και πιο λεπτομερώς αλλά η πρώτη μου εκτίμηση είναι ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι προφανές. Υπάρχει ένα gentleman's agreement, μια συμφωνία κυρίων σύμφωνα με τον οποίο από πλευρά σε δημοσίου δικαίου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν είναι δεσμευτική αλλά υπάρχει και το παράδογο δίκαιο και η θέση του Συμβουλίου είναι στη μέση. Αγγλικά είναι ανακοίνωση, communication ε, ενώ ε, γερμανικά είναι υπόμνημα και θεωρώ ότι είναι μία υποχρέωση νομική αλλά πρέπει να δούμε μέχρι ποιου σημείου φτάνει και αν ε, όντως αυτό ισχύει μόνο για την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ή και για τις Επιτροπές. Θα το ψάξω και θα σας πω. Όσον αφορά τον έλεγχο της νομιμότητος αυτό δεν μπορεί να σημαίνει όπως είπα και στην ομιλία μου ότι περιλαμβάνονται και οι αρχές της καταρτήσεως του προϋπολογισμού δηλαδή η οικονομική σκοπιμό της εάν δηλαδή τα, οι δεν συνάδουν με τις άλλες αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού. Να απαντήσω τις ερωτήσεις με τη σειρά που τέθηκαν. Δεν θέλω να προδικάσω τίποτε, θα ήταν ιδιαίτερα Δεν, δεν θέλω εγώ να προδικάσω τίποτε. Κάποιος είπε είναι πολιτικό το ζήτημα και όταν έχουμε μία αμφίσιμη ερμηνεία στις συνθήκες πάντα υπάρχει μία πολιτική απόφαση από πίσω. Όλα εξαρτώνται από την ομολογική πολιτική της, ε, του δικαστηρίου ε, και κανένας δεν μπορεί να την κατηγορήσει γι' αυτό. Υπάρχει ένας κύκλος ε, γύρω από όλο αυτό το θέμα. Ε, πολλές φορές την κατηγόρησαν για πρωτοποριακές αποφάσεις όπου μιλούσαν για κυβέρνηση των δικαστών. Σήμερα βρισκόμαστε σε μία, από το 2000 και μετά σε μία φάση συγκράτησης και οπισθοχώρησης. Είχαμε, ε, ξέρουμε ότι υπάρχει μία ιδιαίτερα ευαίσθητη ε, ερμηνεία ε, για τις ε, χώρες εκείνες οι οποίες, ε, των οποίων το έλλειμμα ξεπερνούσε το όριο των κριτηρίων σύγκλησης και εκεί υπήρχε μια τεράστια αμφισημία στην απόφαση του δικαστηρίου. Προσπάθησε να τα τακτοποιήσει όλα λέγοντας ότι το Συμβούλιο δεν υποχρεούται να ακολουθήσει τις προτάσεις της Κομισιόν αλλά πρέπει να ακολουθήσει τις προτάσεις της σύστασης Δηλαδή προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Τώρα σε περίπτωση μίας προσφυγής ε, τι θα απαντούσε εγώ δεν μπορώ να δεσμευτώ. Για το θέμα της πληροφόρησης θα έδινε δίκιο αν είμαστε σε μια λογική ισορροπία, θα έδινε δίκιο στο κοινοβούλιο αλλά θα για την πληροφόρηση και την απαλλαγή δύσκολα μπορεί κανείς να το μαντέψει παρά τα επιχειρήματα τα οποία τίνουν υπέρ. Θα ήταν υπέρ των κρατών περισσότερο, τώρα θα φάει τόσο μακριά, δεν ξέρουμε. Ε, μια κυρία που έφυγε Ρώτησε αν η Κομισιόν είναι υπεύθυνη καθαρά και εξάστερα. Ε, όχι. Εγώ λέω όχι καθαρά και εξάστερα, διότι υπάρχει μία αμφισημία, ένα τους μεταξύ της ε, ε, συνθήκης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και το παράγωγο δίκαιο. Δεν μπορούμε εμεί να λέμε ότι είναι καθαρά και εξάστερα η Κομισιόν υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και στην πράξη και στο δίκαιο είναι λάθος. Τώρα η νομική, ε, η νομική αξία του εθιμικού ε, τα συνταγματικά δικαστήρια για να προχωρήσουν το διεθνές δίκαιο χρησιμοποιούν αυτήν την έννοια του εθιμικού δικαίου. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το χρησιμοποίησε πολύ λίγο το εθνικό δίκαιο. Χρησιμοποιεί αυτό των κρατών μελών ή του διεθνούς δικαίου, αλλά όταν δεν υπάρχει κείμενο χρησιμοποιεί τις γενικές αρθές του δικαίου. Αν θέλετε εσείς να την παρασύρετε προς αυτόν τον δρόμο του εφημικού, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου. Τώρα αν το Συμβούλιο αρνιόταν να στείλει ε, τα έγγραφα, μα οι επιπτώσεις θα ήταν μηδενικές, δηλαδή θα δαχτυλοδείχναμε το Συμβούλιο, θα, αρνητικές, υπήρχαν αρνητικές αντιδράσεις, αλλά τίποτα το φοβερό. Όπως εξηγούμε όμως εμείς τους ε, φοιτητέ ε, της νομικής, ε, λέμε ναι εντάξει ένα δικαστήριο καταδικάζει ένα κράτος, αλλά μετά τι γίνεται. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Πόσο μάλλον λοιπόν ε, και ε, όταν πρόκειται για το Συμβούλιο της Ένωσης. Τι γίνεται τότε, παίζουμε στο συσχετισμό δυνάμεων, ε, επαναλαμβάνουμε συνέχεια την προσφυγή. Δεν μπορούμε να στείλουμε εμείς όμως στρατό στο Συμβούλιο για να το υποχρεώσουμε να στείλει τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ την καθηγήτρια την κυρία Σάστε, ο καθηγητής Ρώση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με ευγένεια δεχθήκατε την ε, πρότασή μου, ακούσατε την πρότασή μου, την οποία άμα την εξετάσετε εις βάθος, δεν είναι και τόσο διαφορετική στο προς το δικαίωμα πληροφόρησης του Κοινοβουλίου Νομίζω ότι φάνηκε σαφώς η θέση μου. Ο κύριος Σόνεγκαρ ρώτησε ποιες θα ήταν οι πιθανότητες να κερδίσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα είχατε περισσότερες πιθανότητες όμως αν στο δικαστήριο δεν τρέχατε το Συμβούλιο αλλά την Κομισιόν. Τώρα για ένα τόσο ελάχιστο πια ποσοστό του προϋπολογισμού δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν είναι διαθέσιμο να ασκήσει την αμοιβαιότητα. Το Συμβούλιο μπορεί να παρουσιάσει μία σύσταση ως προς την απαλλαγή αυτό προβλέπει η συνθήκη και ορίζει κάποιες αρμοδιότητες. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο δηλαδή να ξεκινήσουμε μια τέτοια μάχη. Και για να απαντήσω σε άλλες, στις υπόλοιπες ερωτήσεις, να απαντήσω και στους συναδέλφους. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πρωτογενές δίκαιο μπορεί να συνδεθεί με την αλλαγή ε, του οικονομικού πλαισίου. Άμα δούμε τι γίνεται από το 1976 και μετά υπάρχει μία δήλωση εκείνη του 1973 όπου το Συμβούλιο έκανε αυτή τη δήλωση γιατί το Κοινοβούλιο δεν είχε δικαιώματα και αρμοδιότητες. Εκείνη η δήλωση πάντως ε, δεν είναι δεσμευτική και δεν έχει αντικείμενο διότι κατά, σε όλες τις φάσεις τροποποίησης της συνθήκης το Συμβούλιο έκανε τα πάντα για να νοθεύσει το ζήτημα. Τώρα, ρωτώ εγώ, ποιες είναι οι επιπτώσεις, δεν υπάρχει μια νομική επίπτωση. Αυτό μπορούμε να το εννοήσουμε ως εξής. Καταρχήν, το κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιπαρατεθεί με την Κομισιόν, όχι με το Συμβούλιο. Στη διαδικασία απαλλαγής μπορεί κάλλιστα το Κοινοβούλιο να παραχωρήσει την απαλλαγή, να κάνει συστάσεις και παρατηρήσεις για γύρω σημεία και όπως είπε και ο δόκτορας Άμπολεχ, Αυτές οι συστάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σχετικά. Τώρα, αν το θέμα του προϋπολογισμού είναι τόσο πια το επινόδες και θέλουμε κάτι ε, παραπάνω και θέλουμε την άρνηση της απαλλαγής, μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε προσφυγή. Η υπόθεση Σαντέρα πέδειξε ότι ο βασικός ε, ενδιαφερόμενος είναι η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε δύο πυλώνες και εδώ ε, ε, δεν συμφωνώ με την ε, καθηγήτρια Σαλτιέλ. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2 αναφέρεται σαφέστατα το Συμβούλιο αποτελεί έναν από τους φέροντες κορμούς της Ένωσης και δεν έχει νόημα να, να, να κάνουμε πόλεμο. Πρέπει να δεχθούμε και να σκεφτούμε και εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τον κύριο Γκάγερ σίγουρα πρέπει να σκεφτούμε που, να, που πολιτικά να μας ευνοεί και αυτή είναι, αυτός είναι, αυτή η σκέψη που πρέπει να κάνετε το άρθρο 335 και ευχαριστώ για αυτήν τη διευκρίνηση το άρθρο 335 έχει μια εντελώς διαφορετική λειτουργία και ε, αποδεσμεύει άλλα θεσμικά όργανα αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος εξαρτάται από την αυτονομία διαφόρων θεσμικών οργάνων και την διαθεσμική ισορροπία ε, αλλά εις ε, τις επόμενες ημέρες ε, θα λάβετε την τελική μου έκθεση γραπτός εγώ έμαθα πολλά από σας θα, θα προσαρμόσω τα επιχειρήματά μου και στα πλαίσια μίας ανοιχτής συζήτησης πιστεύω ότι μου έκανε καλό που συμμετείχα σε αυτή τη συζήτηση συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ. Σχετικά με την ε, παρατήρηση ε, ε, κύριε Ρώση ότι θέλουμε να υπάρχουν αντιπαραθέσεις και δεύτερον χθες ίσως ε, οφείλεται στην ε, ψηφοφορία μας που δεν παρέστη το Συμβούλιο σήμερα αλλά ε, ίσως και όχι και τώρα έχουμε την τοποθέτηση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρακαλώ τον Ρικάρντο Πάσος να παρουσιάσει τα σχόλιά του και στο τέλος θα δώσω για μία τελευταία φορά το λόγο στους συναδέλφους. Ναι. Συζήτηση χωρίς ε, μικρόφωνο. Ο κύριος Πάσος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσατε πολλά νομικά επιχειρήματα. Όταν καλεί κανείς τέσσερις δικηγόρους, αυτό γίνεται. Ξέρετε ποια είναι η δική μου γνώμη για το θέμα εδώ και καιρό. Δεν θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι συμφωνώ με ό,τι έχει κάνει το Κοινοβούλιο μέχρι τώρα γιατί αυτές τις συμβουλές του έδινα εξάλλου. Είμαι σίγουρος όμως ότι χρήσιμο ήταν να ακούσετε και άλλες γνωμοδοτήσεις άλλων νομομαθών. Δεν χρειάζεται να ξανακάνω το ιστορικό. Η κρίση, γιατί κάποιος ανέφερε τη λέξη αυτή, αν υπάρχει κρίση, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει για κρίση. Η διαμάχη, ας πούμε έτσι, από το 2009 ή από την θέση ενισχύ της συνθήκης Λισαβόνας είναι πιο φανερή από πλευράς του Συμβουλίου ως θεσμικού οργάνου, το οποίο δεν είχε θεσμοθετηθεί τόσο επίσημα μέχρι τότε. Το θέμα αφορά τη δημοκρατική νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την απαλλαγή. Ακούστηκαν επιχειρήματα ως προς το κατά το Κοινοβούλιο έχει τη δικαιοδοσία να δίνει χωριστά απαλλαγή για το Συμβούλιο. Εγώ θα περιουστώ σε τρία επιχειρήματα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου έχει αλλάξει. Το είπε κάποιος. Στην αρχή μόνο το Συμβούλιο είχε δικαίωμα να δίνει απαλλαγή και από το 70 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και τώρα μετά από το 75 τη συνθήκη των Βρυξελών μόνο το Κοινοβούλιο δίνει απαλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια εξέλιξη στο ρόλο του Κοινοβουλίου ως προς την απαλλαγή. Τα τρία σημεία που ήθελα να τονίσω είναι φυσικά υπέρ της απαλλαγής, χωριστής απαλλαγής για το Συμβούλιο. Όχι όμως με βάση με μονομένα άρθρα της συνθήκης αλλά με το συνδυασμό τους. Το δεύτερο επιχείρημα αφορά το παράγωγο δίκαιο που δίνει δικαίωμα σε χωριστή απαλλαγή και το τρίτο είναι το επιχείρημα της απαλλαγής ως τμήματος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, διαφάνειας και καλής διακυβέρνησης. Το πρώτο στοιχείο για το 319 Στις παρουσιάσεις που έγιναν, με όλο το σεβασμό που οφείλω στους εισηγητάς και ιδίως τον καθηγητή Ρώση, θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μια κυριολεκτική μόνο ερμηνεία του 319 το οποίο πράγματι αναφέρει ρητά ότι το Συμβούλιο δίνει απαλλαγή στην Κομισιόν. Ναι, αλλά πρέπει να διαβάσουμε όλη τη φράση που λέει εξή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σύσταση από το Συμβούλιο δίνει απαλλαγή στην Κομισιόν ως προς την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Αυτή η φράση ως προς την, απαλλαγή του ως προς την εφαρμογή του προϋπολογισμού είναι σημαντική διότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι κάτι που έχει ερμηνευθεί και εξελιχθεί. Και δεν πρέπει να περιοριστούμε στη λέξη κομισιόν εδώ. Επίσης, εκτέλεση του προϋπολογισμού πρέπει να ξέρουμε ότι γίνεται μόνο κατά 10% από την Κομισιόν άμεσα. Άρα, όπως είπε η κυρία Γκρέσλε, έχουν αλλάξει τα πράγματα από η Κομισιόν είναι άμεσα υπεύθυνη μόνο για το 10% της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Υπάρχουν και τα άλλα όργανα που τον εκτελούν. Αυτό το μέρος λοιπόν του 319, αν και για μερικούς θεωρείται σαφές, δεν μπορεί να ερμηνευτεί μόνο κυριολεκτικά. Γιατί πρέπει να συνδυαστεί και με το 317.2. Και τι λέει το 317.2? Το 317.2 λέει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός καθορίζει τις ευθύνες και δικαιοδοσίες για κάθε όργανο για τη δαπάνηση του υπολογισμού του. Αυτό σημαίνει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός μιλάει ρητά για χωριστές απαλλαγές. Υπάρχει το άρθρο 50 του που λέει ότι η Κομισιόν συνεννοείται με, ε, χορηγεί στα άλλα όργανα τις δικαιοδοσίες εκτέλεσης του προπολογισμού τους. Το 146 παράγραφος 2 λέει επίσης ρητά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη χορήγηση της απαλλαγής εξετάζει την ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και τις απαντήσεις που έχουν δώσει τα άλλα όργανα και το 147 λέει ότι η Κομισιόν και τα άλλα όργανα θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να ακολουθηθούν οι συστάσεις που θα αναφέρονται στην απαλλαγή του Κοινοβουλίου, από το Κοινοβούλιο. Όλα αυτά του δίνουν, του Κοινοβουλίου, σταθερή βάση να συνεχίσει τα πράγματα όπως το έπρατε μέχρι τώρα με χωριστές απαλλαγές. Και τελευταίο επιχείρημα, το τρίτο, πιο ουσιώδες και δεν έχει ακουστεί και τόσο πολύ. Αφορά και τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπως το ανέφεραν οι ομιλητές. Η θέση του Κοινοβουλίου άλλαξε μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ζούμε σε κράτος δικαίου το οποίο βασίζεται στην αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο ανοιχτά και διαφανώς γίνεται. Άρθρο 10 παράγραφος 3. Επίσης όμως συνδέεται με αυτό άλλο άρθρο της συνθήκης η αρχή της καλής διακυβέρνησης και αυτό το 15.1 απαιτεί για να προωθηθεί καλή διακυβέρνηση τα ενωσιακά όργανα να λειτουργούν όσο δυνατόν πιο ανοιχτά. Τώρα για θέματα του προπολογισμού και της εκτέλεσής του υπάρχει η αρχή της διαφάνειας στον δημοσιονομικό κανονισμό 29, το άρθρο 29 τώρα 31 προβλέπει ο προϋπολογισμός να εκτελείται με βάση την αρχή αυτή. Αυτές τις βασικές αρχές λοιπόν της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τις συνδυάσουμε με το δημοσιονομικό κανονισμό, δίνεται νέα διάσταση στην ερμηνεία του 319 και στο ρόλο του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή. Πρέπει επίση να πούμε σε αυτά τα πλαίσια ότι πρόκειται για δημόσιο χρήμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέδειξε ιδιαίτερη αυστηρότητα ως προς αυτό και αναγνώρισε ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα δημόσια χρήματα. Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και τέτοιος έλεγχος δεν μπορεί να γίνει, συμφωνώ εδώ με την καθηγήτρια Σαλτιέλη, παρά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι το μόνο όργανο που είναι άμεσα εκλεγμένο από τους πολίτες. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ να τελειώσω εδώ. Ακούσαμε επιχειρήματα που στηρίζουν τη θέση του Κοινοβουλίου. Και θα σταματήσω εδώ για πληροφόρηση των νομικών εμπειροχνωμόνων που ίσως δεν το γνωρίζουν, θα ήθελα να πω ότι η θέση του Κοινοβουλίου για χωριστές απαλλαγές έχει γίνει δεκτή από όλα τα θεσμικά όργανα, εκτός από το Συμβούλιο. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής εδώ έχει στείλει επιστολή στον αρμόδιο επίτροπο, όπου του ζήτησε, το ρώτησε, ποια είναι η θέση της Κομισιόν. Και ο Επίτροπος Σίμηταρ πριν από λίγο καιρό, τον Νοέμβριο του 2011, απάντησε ότι η Κομισιόν γνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στα άλλα όργανα χωριστά για πολλά χρόνια και ότι ποτέ δεν αφισβητήθηκε η διαδικασία αυτή από την Κομισιόν, την θεωρεί δε θεμητή και στο μέλλον θα συνεχί... ότι πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται έτσι. Αυτό το αναφέρω διότι θέλω να απαντήσω και στα επιχειρήματα που ανέφεραν ορισμένοι ότι δηλαδή όλα πρέπει να περνούν από την Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει περιορισμένη ευθύνη για την εκτέλεση του προπολογισμού. Πρόεδρε, καταλήγω, αν μου το επιτρέπετε, απαντώντας στα τρία ερωτήματα που τέθηκαν στους εμπειρογνώμους. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να πω τίποτα ως προς το κατά πόσον είναι ευχή έργων να γίνει προσφυγή από το κοινοβούλιο στο δικαστήριο. Κατανοείτε γιατί κολλείομαι να το κάνω αυτό. Είναι θέμα που πρέπει ακόμη να συζητηθεί, αλλά όχι σε αυτό το βήμα. Θα είμαι σύντομος για τα άλλα. Πρώτον, κατά πόσον υπάρχει η οθός. Δεν συμφωνώ εδώ με την καθηγήτρια Σαλτιέλ. Νομίζω ότι εδώ υπερβάλλει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει εδώ ήθος ή ιωθός για αυτό το θέμα της απαλλαγής. Γιατί είναι όρος πολύ γνωστός και πολύ ισχυρός στο διεθνές δικαίωμα και δεν αφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, κατά πόσον αυτή η συμφωνία κυρίων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου είναι νομικά δεσμευτική. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα αυτό γιατί για ένα πολύ απλό λόγο η συμφωνία κυρίων δεν αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού καθόλου αλλά μόνο τον καθορισμό του όχι την εφαρμογή του, την εκτέλεσή του. Κατά πόσο λοιπόν είναι νομικά δεσμευτική ή όχι είναι άλλο θέμα. Εγώ τίνω να πιστεύω ότι οι συμφωνίες κυρίων είναι νομικά δεσμευτικές αν συμφωνούν και τα δύο μέρη. Ίσως λοιπόν να είναι νομικά δεσμευτική αλλά όχι ως προς την απαλλαγή. Τέλος. Για τις συνέπειες της απαλλαγής εδώ συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε ότι δηλαδή δεν υπάρχουν νομικές επιπτώσεις για την άρνηση της απαλλαγής. Οι επιπτώσεις είναι πολιτικές. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Πάσος για τη σημαντική σας συμβολή και τώρα αρχίζει η γενική συζήτηση ή αν θέλετε και άλλες ερωτήσεις για τους εμπειρογνώμονες. ανάλογα με το χρόνο θα δω αν υπάρχει δυνατότητα για καμιά συντομή απάντηση. Πρώτα η συγγήτρια κυρία Γιάλα Σέντερ. Εγώ πρόεδρε απλώς ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στον κύριο Ρώση Ε, για το θέμα του, της ιστοσελίδας πέρα από την ιστοσελίδα των, φιλελευθέρων που σας θυμά, κύριε Πρόεδρε δεν έχει παρά και να κοιτάξει και την ιστοσελίδα ε, της σοσιαλιστικής ομάδας. Ε, με σοκάρισε αυτό. Γιατί δηλαδή μόνο το, την ιστοσελίδα τη ομάδα των φιλελευθέρων. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, όλο το υλικό και όλα τα έγγραφα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Κυρία Γέσλερ. Έχω μία ερώτηση στον καθηγητή Ρώση για την αμοιβαιότητα αρνηθήκαμε αυτή την αμοιβαιότητα γιατί δεν υπάρχει ισοτιμία, equal footing, αλλά το Συμβούλιο δίνει μία σύσταση. Εάν συνδυάσουμε τη σύσταση με την απαλλαγή, ε, δίνει ε, κανονικά για τους κανονισμούς συστάσεις στο Συμβούλιο. Μπορεί να θεωρηθεί ισότιμη, η ισότιμη ε, ε, η ισότιμη απαλλαγή από το Συμβούλιο, η απαλλαγή από το Κοινοβούλιο με τη σύσταση του Συμβουλίου ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Επίσης υπάρχει εδώ ένας πίνακας στον οποίο καταρτήσαμε με τροπολογίες στην απαλλαγή για να τονίσουμε ε, πώς έχει εξελιχθεί η νομική θέση. Υπάρχει, υπάρχουν ε, τροπολογίες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ε, υπάρχει δηλαδή μία συνεχής κατάσταση που πρέπει να εξελίσσεται και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους στις τις εργασίε ε, για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαίου να περιλάβουν αυτή την πτυχή γιατί βρίσκω ότι η ε, γερμανική νομολογία δεν προωθεί την ε, ευρωπαϊκή. Ε, πρέπει να καταστήσουμε πιο συγκεκριμένα τα θέματα που παρουσιάσουμε εδώ. Άκουσα προσεκτικά και αυτό που είναι βασικό είναι το δίκαιο να μπορέσει να αναπτυχθεί μαζί με τους προβληματισμούς και το Συμβούλιο επίσης από κοντά. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να παρέμβει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε κύριε Ρώση, εσείς ε, ε, ε, θεωρήσατε ότι η Γερμανία είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος και υπάρχει με μεταξύ του Bundestag και Bundesrat του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και της Γερουσίας και το Συμβούλιο έχει την αυτονομία και ε, τον προϋπολογισμό αλλά ε, το Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά του Bundesrat της Γερμανικής Γερουσίας ε, ως προς τις, τα δημοσιονομικά θέματα και το ερώτημα είναι, έχουμε τις ίδιες δυνατότητα και το άλλο μπορεί κανείς να το εξασκήσει όντως, δηλαδή στην πρακτική τι γίνεται. Επ' αυτού θα ήθελα να μου σχολιάσετε και να μου πείτε πώς βλέπετε ε, τη ε, συγκρισιμότητα ε, ότι ένα άλλο θέμα που ανέφερε ο συνάδελφός σας είναι ότι η θα μπορούσε ε, το Συμβούλιο να ελεγχθεί από τα εθνικά κοινοβούλια ε, στην Γερμανία υπάρχουν και τα, ε, και τα κοινοβούλια των κρατηδίων και το Bundestag και τα κοινοβούλια των κρατηδίων δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τον Bundesrat στη Γερουσία δηλαδή και ε, εάν ε, ε, υποθετικά προβεί κανεί αυτή τη σύγκριση είναι σαν να πούμε ότι θεωρητικά χτίζουμε ένα νέο αεροδρόμιο υπάρχουν έξοδα και υπερημερίες και μπορεί το κοινοβούλιο να επέμβει ενώ εδώ εάν υπάρχουν καθυστερήσεις σε παράδοση κτηρίων το ερώτημα είναι ποιος ε, είναι υπεύθυνος ε, αυτό μπορεί να προκύψει και για την ε, ελεγκτική αρχή και δεν ήταν τυχαία τα δείγματα που ανέφερα και μπορείτε να σχολιάσετε σαν, σαν νομική. δεν κατάλαβα την παρατήρηση της ομιλήτριας. Ίσως υπάρχει μία παρανόηση ίσως ε, ε, ε, εγώ προσπάθησα να είμαι αντικειμενικός από πλευράς πολιτικής σαν επιστήμονας. Δεύτερον, το θέμα της αμοιβαιότητος. Δεν συμφωνώ μαζί σας διότι όντως, δηλαδή δεν, δεν πρόκειται για υποχώρηση, είναι μία βάση. Μία σύσταση είναι μία σύσταση και όταν το, θέλετε να μην δώσετε απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορείτε να το πράξετε. Εάν όμως δεν θέλετε να απαλλάξετε το Συμβούλιο διότι ε, το Κοινοβούλιο ε, δεν έχει ε, σεβαστεί τις υποχρεώσεις τους τότε το Συμβούλιο πρέπει να μπορεί να επέμβει επί του συγκεκριμένου θέματος. Άρα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότης διότι διαφορετικά υπάρχει ένα σχεδόν θεωρητικό θέμα ποιος παρακολουθεί ε, τους ε, παρατηρητές και φαντάζομαι ότι σε αυτό το σημείο δεν θα συμφωνήσουν όλοι οι συναδελφοί σας και τι προβάλλει αυτό προς τα έξω. Δηλαδή χρειάζεται ενημέρωση διότι όντως υπάρχει κοινή αντιμετώπιση διότι το ελεγκτικό συνέδριο έχει και αυτό αρμοδιότητες και αυτό θα αξιολογήσει την έλλειψη της τοποθέτησης του Συμβουλίου όσον αφορά τις σχέσεις ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ο επιεθνικού, γερμανικού και ευρωπαϊκού επίπεδου νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ότι ε, μία ομοσπονδιακή δομή ε, μπορεί να βοηθήσει σε μία σύγκριση ακόμη και αν δεν είναι απολύτως ταυτόσιμη. Ε, στην αρχή ε, ε, ε, έκανα την σύγκριση αυτή και είχα αντιληφθεί ότι το ερώτημα ήταν εάν το Bundestag μπορεί να αρνηθεί την απαλλαγή στο Bundesrat και επί του προκειμένου πιστεύω ότι όπως και στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι αυτό επιτρεπτό και η υπεύθυνο ε, και αποδέκτης της απαλλαγής είναι η κυβέρνηση όπως εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν έκανε ίσως καλά τη δουλειά της και το Bundesrat πέραν ε, των δογματικών ε, διαφορών δεν είναι καλό παράδειγμα διότι δεν έχει καμία εκτελεστική, ε, εκτελεστική εξουσία και μειώθηκε ό,τι είχε από την Λισαβόνα. Δεν έχω τώρα τους αριθμούς αλλά ο όγκος του Συμβουλίου είναι χαμηλότερος τώρα αλλά πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να συλλέξει τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται ε, για τον προϋπολογισμό από ε, το Bundesrat και από το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ε, είπατε κι εσείς και εγώ το ανέφερα επίσης ότι δεν μπορεί κανείς να εμπλέξει τα εθνικά κοινοβούλια στη διαδικασία απαλλαγής του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει εθνικός κατακαιρματισμός και συμφωνώ με τους συναδέλφους ε, διότι το Κοινοβούλιο δεν είναι εποπτική αρχή και όσον αφορά ε, τις νομικές δυνατότητες ας μην έχουμε ψευδευσίσεις δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει έναν υπουργό να παρετηθεί γιατί δεν εκτέλεσε ε, σωστά τον το, τμήμα του προπολογισμού που του αναφέρεται. Ε, είσαστε όμως επαγγελματίας και ξέρετε ότι ένα ένα θέμα το οποίο έχει επί εβδομάδες πολιτικές επιπτώσεις δεν μπορεί να καθυστερεί. Ευχαριστώ. Ο άλλος Ε, αναφέρθηκα στη σελίδα ε, αναφέρθηκα στο θέμα της αμοιβαιότητας και εγώ όπου συμφωνώ σχετικά με την ε, πρόταση Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί να υπάρξει πρόταση, δεν υπάρχει πλήρης αμοιβαιότης και το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα πληρεφόρησης διότι ε, μπορεί στο άρθρο 319 παράγραφος 1 αναφέρεται και το Κοινοβούλιο και ε, το Συμβούλιο ενώ στην παράγραφο 2 αναφέρεται μόνο το Κοινοβούλιο και όχι το Συμβούλιο και αυτό ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο και στον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν υπάρχει αμοιβαιότηξη μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και δεν είναι προφανές εάν οι πληροφορίες που λαμβάνει το Κοινοβούλιο πρέπει να παραπέμπονται και στο Συμβούλιο στην ισότιμη συνεργασία αλλά δεν είναι τα δικαιώματα τα ίδια μεταξύ των δύο. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαλέλα δεν ζητά τον λόγο και θέλω να δώσω τέλος το λόγο στην εισηγήτρια Γιάλα Σέντερ εάν το επιθυμεί. Ε, ευχαριστώ. Λυπούμε για το, για το, για το web, ε, έκανα λάθος ε, εγώ, διότι στο κείμενο η κυρία Σαλτιέλ είναι αυτή που συμβουλεύθηκε το, την ιστοσελίδα των φιλελευθέρων και όχι ο κύριος Ρώση, αλλά δεν φαινόταν επί του κειμένου. Λοιπόν, συμβουλεύω τότε την κυρία Σαλτιέλ να συμβουλευτεί άτρες ιστοσελίδες. Ήταν πολύ καλή ιδέα αυτό το σεμινάριο. Βέβαια το Συμβούλιο θεώρησε ότι δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα να έρθει εδώ να εξηγηθεί και πιστεύω ότι δεν είναι μια καλή στρατηγική το να αποφεύγουν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα την ε, δημόσια συζήτηση, το γιατί, για τις δράσεις τους ή όχι. Εγώ καταλαβαίνω ε, στην ευρωπαϊκή στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχουμε στοιχεία νοριμότητας. Αυτό είναι και η δημοκρατικότητα. Εμείς έχουμε εκλεγεί εδώ οι ευρωβουλευτές σε εθνικό επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό. Αλλά η νομιμότητα του, ε, η δημοκρατική νομιμότητα του Συμβουλίου σίγουρα είναι δημοκρατική νομιμότητα σε επίπεδο επίπεδο των εθνικών του κοινοβουλίου δεν είναι για να υπόλογο για τις δαπάνες του και τα έξοδα του έναντι του μοναδικού οργάνου που έχει δημοκρατικά εκλεγεί και που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκκρεμεί ακόμη η συζήτηση. Πρόκειται για μία ε, αρχή η οποία ακόμη βρίσκεται σε... που είναι καθαρά πολιτική έστω και αν έχει ακόμα ακαδημαϊκό χαρακτήρα θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα την επόμενη εβδομάδα που θα συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό και σε αυτήν την μάχη η ευθύνη του Συμβουλίου έναντι του Κοινοβουλίου και για το θέμα δηλαδή της απαλλαγής θα πρόκειται για ένα παράπλευρη ζημιά. Και θα είναι μια ζημιά παραπάνω. Τώρα εγώ από τη μέρα που μπήκα σε αυτό το κοινοβούλιο το 1997, τότε ο Κεν Κόλινς μου είχε δώσει και το πρώτο μάθημα ήταν πρόεδρος της Επιτροπής, ε, ε, της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και τότε εγώ ως υπάλληλο της ομάδας τον είχα, του είχα ρωτήσει δεν είναι γραμμένο κύριε πρόεδρε και μου απάντησε ακριβώς επειδή δεν είναι γραμμένο γι' αυτό θα το παλέψουμε. Εμείς θα το παλέψουμε λοιπόν όπως κάνουμε κάθε χρόνο, σχολιάζει το ελεγκτικό συνέδριο, το, κοινοβου... Συμβούλιο δέχεται αυτά τα σχόλια και μετά τα σχολιάζει. Και μετά δίνεται και η απαλλαγή. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε δίκιο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο με τις προτάσεις της κυρίας Σαλτιέλ είτε με πίεση της κοινή γνώμης, ε, ε, η πίεση των ε, ΜΜΕ και τέλος πάντων επειδή θα αποφασίσει το Συμβούλιο ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και δεν θα αμφισβητεί και τη δική μας νομιμότητα τότε θα δεχθεί να υποκύψει το Συμβούλιο έστω και αν πρόκειται για ένα ελάχιστο τμήμα του προϋπολογισμού ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ξέρει που ξοδεύονται τα λεφτά του. Αυτά κύριε Πρόεδρε, εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι την Ολομέλεια. Εδώ πρόκειται για μια περαιτέρω φάση. Ε, ήταν μια ευκαιρία να έρθει το Συμβούλιο να εξηγηθεί, αλλά δεν ήρθε. Εμείς θα συνεχίσουμε να τους ε, καλούμε και να έρθουν και στην Ολομέλεια και λοιπά για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια Γιάλα Σέντερ για αυτές τις ε, παρατηρήσεις ε, που συνόψισαν τη συζήτηση. Ψάχνουμε να βρούμε μία επικοδομητική λύση και αυτό είναι κάτι που θέλω να τονίσω και όσον αφορά τις παρατηρήσεις σας κύριε Ρώση ότι το Συμβούλιο ίσως ε, χρειάζεται ε, πληροφορίες από το Κοινοβούλιο για να ολοκληρώσει τη θέση του δεν έχουμε πρόβλημα και δεν αντιτιθέμεθα ε, εμείς προσπαθούμε ε, τα στοιχεία του Συμβουλίου να διατίθενται με πλήρη διαφάνεια εις το διαδίκτυο κατά τρόπον ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια για τη σωστή χρησιμοποίηση των πόρων και των οικονομικών των φορολογουμένων. Η απαλλαγή είναι δικαίωμα του Κοινοβουλίου και όχι μόνο αυτής της Επιτροπής που προβαίνει στις προκαταρκτικές ε, παρατηρήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, νομικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι μας επέτρεψαν μια καλύτερη ερμηνεία των ε, συνθήκων τον κύριο Ρώση, τον κύριο Εντβέλερ, την κυρία Σαλτιέλ και σας ευχαριστώ που συμμετείχατε εδώ. Φαντάζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε προχωρήσει για την ε, περαιτέρω πρόοδό μας και ο στόχος τον οποίων επιζητούμε είναι να υπάρχει ο πλέον δημοκρατικός έλεγχος. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία και το Policy Department και τον κύριο Φίσερ για την πρωτοβουλία και Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τους εξωτερικούς ε, ε, συνεργάτες μας, ε, τους φιλοξενούμενους μας, να τους δώσω από ένα βιβλίο για 50 χρόνια ιστορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μην μας ξεχνάσουν. Επίσης ε, ε, έχουμε έναν συνάδελφο ο, ο οποίος φεύγει από τη γραμματεία μας και μεταφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θέλω να του πω ότι μας έχει διευκολύνει μέχρι σήμερα τη δουλειά και εύχομαι να τον ξαναδούμε σύντομα.